Bitte nehmen Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Για καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Ich heiße alle herzlich willkommen hier heute. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας συνεδρία του 2011 και επειδή είναι και η πρώτη μας ε, συνεδρίαση, σας εύχομαι καλό 2011 με χαρά, με υγεία, με επιτυχία. Ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό, να είναι έτος υγείας, χαράς και επιτυχίας και να λειτουργήσουμε και να εργαστούμε σωστά. Πέναμε στην σε διάταξη αμέσως γιατί το θέμα μας σήμερα είναι η μελλοντική αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαμόρφωσή της και η χρηματοδότησή της. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον Επίτροπο κύριο Τσόλος μαζί μας, ο οποίος είναι έτοιμος να ανταλλάξει απόψεις μαζί μας και να μας εξηγήσει ποια είναι τα σχέδια της Κομισιόν σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος του κυρίου Επιτρόπου. Δεν θα μπορέσει να μείνει μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασής μας. Θέλω λοιπόν να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι θα αλλάξω, δεν μου έρχεται η γερμανική λέξη, βέξεν, θα ανταλλάξω τα σημεία 3 και 4 Λοιπόν, ελπίζω να συμφωνείτε λοιπόν να αλλάξουμε τη σειρά των σημείων 3 και 4. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να σας ανακοινώσω, αλλά δεν είναι πρόβλημα να το κάνω στη συνέχεια όταν έχουμε συζητήσει ήδη με τον κύριο Επίτροπο. Θα περάσουμε λοιπόν πρώτα στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης Αν δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντίρρηση για τα πρακτικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Αν μέχρι το τέλο τη συνεδρία δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Σημείο λοιπόν 4 τη ημερήσια διάταξη. Μελλοντική αγροτική πολιτική μετά το 2013, γιατί μέχρι το 2013 είναι ρυθμισμένα όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς θέλουμε να αλλάξουμε την κοινή αγροτική πολιτική επέκεινα του 2013 και ποιες θα είναι οι συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μπούμε τώρα στην εργασία της επεξεργασίας των μελλοντικών αυτών προοπτικών. Θα δώσω λοιπόν στο Σαλβαδόρ το λόγο για 5 λεπτά και μετά στην Κομισιόν για 10 λεπτά για να εκθέσει τη θέση της Κομισιόν και ενδεχομένω να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί κάποιες από τις οποίες και εγγράφος και ακολουθούν οι ομιλητές εξονομώσεις των πολιτικών ομάδων, όχι κατά ανάγκη οι συντονιστές. Κάποιες ομάδες είπαν ότι θέλει να λάβει το λόγο εξ ονόματός τους κάποιος άλλος από τους συντονιστές. Εν πάση περιπτώσει, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων πέντε λεπτά το maximum ο καθένας. Αν μπορούν να είναι πιο σύντομοι, τόσο το βελτιστότερον. Και θέλω να χαιρετήσω επίσης εδώ και τους εκπροσώπους της Επιτροπής Γεωργίας στη συνεδρίασή μας, που μπορούν να παρουσιάσουν και τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας μετά από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και μετά θα αρχίσει ο πρώτος γύρος απαντήσεων από τον κύριο Επίτροπο και μετά θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και έχουμε ήδη αρχίσει να καταγράφουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο στον επόμενο γύρο με επικεφαλή τον Τζόνι Βαν Λαβία αλλά ξεκινάμε τώρα με τον Σαλβαδόρ Γαρίγα σε παρακαλώ να λάβεις το λόγο Σαλβαδόρ σε ευχαριστώ. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Δεν ξέρω πού είσαστε, αλλά κάπου εδώ είσαστε. Είναι λίγο πίσω στο Σαλβαδόρ. Ναι, ναι, το είχα καταλάβει ότι ήταν κοντά μου. Όπως είπαμε χθες μεταξύ συντονιστών, κυρία Πρόεδρε, το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης, να ακούσουμε τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων για το τι θα πρέπει να πράξουμε με την κοινή αγροτική πολιτική μέσα στα πλαίσια των επερχομένων δημοσιονομικών προοπτικών. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να ακούσω περισσότερο τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Υπάρχουν κάποια πρώτερα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να θέσω στον κύριο Επίτροπο και φυσικά καταρχήν να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του. Νομίζω ότι όπως και πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτημένη αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βρίσκεται και στην πηγή, στην ε, βάση μάλλον της ε, ανακοίνωσης της ε, Κομισιόν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική η ανάγκη όμως αυτή να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική η οποία θα είναι καλά διαμορφωμένη και χρηματοδοτημένη έρχεται σε σύγκρουση με κάποιες ε, δηλώσεις που ακούμε από ορισμένα κράτη-μέλη που πριτανεύουν υπέρ μια συνολικής μείωσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θέλω να θέσω στον Επίτροπο κ. Σόλος είναι ποια είναι η δική του στάση σε σχέση με το συνολικό όγκο του προϋπολογισμού που θα πρέπει να αποδοθεί στην κοινή αγροτική πολιτική ξεκινώντας από το 2013. Θεωρεί δηλαδή ο κύριος ε, Επίτροπος ότι είναι επαρκή τα τωρινά κονδύλια του προϋπολογισμού θεωρεί ότι με τον προϋπολογισμό που επιζητούν ορισμένα κράτη-μέλη που θέλουν να μειώσουν γενικά την ε, χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής ότι θα μπορεί να συνεχίσει αυτή η πολιτική στο μέλλον. Και επίσης πρέπει να έρθουμε και στο υπόδειγμα χρηματοδότησης της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής με τις άμεσες πληρωμές στον πρώτο πυλώνα και τη συγχρηματοδότηση στο δεύτερο πυλώνα. Και εδώ το ερώτημά μου θα συνδεθεί στην απάντηση που θα δώσει ο κύριος Επίτροπος στο πρώτο μου ερώτημα. Θεωρείτε ότι μια πλήρης ε, κοινοτικοποίηση της χρηματοδότησης της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής θα βελτιώσει την απόδοση της πολιτικής ή θέλετε να επεκτείνετε τη χρηματοδότηση και στον πρώτο πυλώνα και όχι μόνο στο δεύτερο. Και όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται <clears throat> από τον όγκο των κονδυλίων, αλλά φυσικά θα πρέπει πέραν αυτού να σκεφτούμε πώς θα ενσωματωθεί η κοινή αγροτική πολιτική σε μια μελλοντική διάρθρωση των δημοσιονομικών προοπτικών. Ξέρουν οι συνάδελφοι ότι εμείς έχουμε παρουσιάσει μια σειρά από επιλογές σε ένα έγγραφο εργασίας που ξεκινά από ένα απλό σύστημα μέχρι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πλέγμα ε, πολιτικών Πρέπει όμως να ευθυγραμμίσουμε σε κάποιο βαθμό την κοινή αγροτική πολιτική με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και αν πράγματι το θέλουμε αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν η γεωργία πρέπει να παραμείνει ως μία αυτόνομη πολιτική ή αν θα πρέπει να κατανεμηθεί στους διάφορους στόχους της ανάπτυξης, της εφηού και αηφόρου ανάπτυξης ή της περιεκτικότητας και της συμπερίληψης και να μην παραμείνει μια αυτόνομη πολιτική. Επίσης παραμένει το ερώτημα του τι θα κάνουμε με το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ορισμένοι θεωρούν ότι όλα τα διάφορα ταμεία θα πρέπει να συνενωθούν <clears throat> υπό την αιγίδα της πολιτικής συμπερίληψης, περιλαμβάνοντας και το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. <clears throat> Αυτή είναι μια επιλογή βέβαια που έχει και τα θετικά και τα αρνητικά της. Θα ήθελα και σήμερα να ακούσω από τα χείλη του κυρίου Επιτρόπου ποια είναι η άποψή του για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι ήμουν πολύ σύντομο, κυρία Πρόεδρε, και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι θα έχουν να θέσουν πιο λεπτομεριακά από μένα ερωτήματα στον κύριο Επίτροπο. Vielen Dank, vielen Dank, Salvatore. Ja, sehr präzise, sehr ähm, äh, gut kurz. Ε, ε, ε, Merci, Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά. Μια χρονιά πλούσια σε καλές ιδέες και εργασίες για το καλό της Ευρώπης. Από την πλευρά μας, από την πλευρά της Επιτροπής, προσπαθούμε και εμείς να εξεύρουμε καλές ιδέες. Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχαμε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και θα περάσω απευθείας στην ουσία. Η ανακοίνωση αυτή στόχο έχει να ετοιμάσει την κοινή αγροτική πολιτική με προοπτική το 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά πρώτον τα όσα ορίζει η συνθήκη, οι, τις αρμοδιότητες που Προβλέπει δηλαδή τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσει και του στόχου η κοινή αγροτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τι ανάγκε τη κοινωνία μα, τι προσδοκίε των πολιτών για τα ερχόμενα χρόνια, μεσοπρόθεσμα. Η κοινή αγροτική πολιτική δεν θα είναι μόνο μια τομεακή πολιτική, αλλά θα έχει διατομεακή εμβέλεια και διαφορετικού ρόλου. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι στόχοι για το μέλλον για την κοινή αγροτική πολιτική. Πρώτα απ' όλα επιστημιστική ασφάλεια. Επιστημιστική ασφάλεια που αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και την ποικιλία των ε, τροφίμων, καθώ και την ασφάλεια. Αυτό βλέπουμε να δείτε το θέμα και από τα δημοσιεύματα του τύπου τις τελευταίες ημέρες. Ε, είναι ένας στόχος που θα πρέπει συστηματικά να επιδιώκουμε και για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα δεύτερο σημαντικό στόχο. ε, όλο και περισσότερο σημαντικό για την ε, κοινή αγροτική πολιτική, είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων και για την οικονομική ζωή, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε του πόρου που μα επιτρέπουν να παράγουμε τρόφιμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στόχο από άποψη ε, οικονομικής αλλά και άποψης περιβαλλοντική. Πρέπει να διασφαλίσουμε την διατηρήση τη βιοπικιλότητας, την ποιότητα των εδαφών, των υδάτων και σε αυτού του στόχου πρέπει να ανταποκρίνεται η γεωργία. Πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά του φυσικού πόρου. Επίση, η γεωργία από κοινού με την δασοκομεία, γιατί εδώ μα απασχολεί και το μέσο των δασών, καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα τη επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό στόχο για την Ευρώπη των 27, που έχει και μεγάλη ποικιλία ω προ τα εδάφη τη, είναι η συμβολή τη Γεωργία, η συμβολή που οφείλει να έχει η Γεωργία στη διατήρηση τη εδαφική ισορροπία και τη ε, ισορροπίας της υπαίθρου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, αυτή η συνοχή θα επιτευχθεί όχι μόνο μέσω τη κοινή αγροτική πολιτική, διότι η κοινή αγροτική πολιτική οφείλει να επιδιώκει συστηματικά το στόχο αυτό, για τον επιπλέον λόγο ότι μετά τη διεύρυνση το θέμα τη υπαίθρου, το θέμα τη εδαφική ακαιρεότητα είναι ακόμα πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, με τη μελέτη που έγινε πρόσφατα, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει και η νέα αγροτική πολιτική να έχει και μια σαφή προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Διότι πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο για πολιτικές που έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η κοινή αγροτική πολιτική λοιπόν είναι πλέον ε, κοινοτική από αυτέ που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική που έχει περάσει από πολλέ μεταρρυθμίσει τα τελευταία έτη και είναι μια πολιτική που έχει να ανταποκριθεί σε οικονομικές αλλά και εδαφικές προκλήσεις. Εδώ μιλάμε λοιπόν για νέα αγορά, αλλά πρέπει να μιλάμε και για διαχείριση όλων των εδαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σαφώς ότι οι πολιτικές σε κοινοτικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές από το να έχουμε 27 εθνικές διαφορετικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν ο προσανατολισμός της μεταρρύθμισής μας ε, λαμβάνει υπόψη οικονομικές προκλήσεις, περιβαλλοντικές, εδαφικές που καλύπτονται και από τη στρατηγική του 2020. Εδώ η κοινή ασματική πολιτική πρέπει να επιδιώκει στόχους ε, όπως προβλέπονται από τη συνθήκη, αλλά και στόχους όπως προβλέπονται από αυτή τη στρατηγική, τη στρατηγική του 2020. Διότι η βιώσιμη διαχείριση δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αύξηση και η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς οικονομική δραστηριότητα γεωργική που να έχει σχέση ακριβώς με την ουσία της γεωργίας. Και η ευφυής ανάπτυξη δεν μπορεί να λάβει χώρα ε, στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων όπου σας θυμίζω ότι η βιομηχανία έχει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών από όλες τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, από όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και εξασφαλίζει τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Σε αυτόν λοιπόν τον τομέα δεν μπορούμε να πετύχουμε θη ανάπτυξη χωρίς εξυγχρονισμό και αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο αγροτικό ε, επίπεδο. Ο τομέα τη γεωργία και των τροφίμων είναι πολύ ισχυρό γιατί ακριβώ η κοινή αγροτική πολιτική μα στηρίζει τον τομέα αυτό και στην ε, διαχείριση, την αποτελεσματική διαχείριση των πρώτων υλών. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτού του στόχου και για να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Γκαρίγκα Πολέδο, προβλέψαμε στόχους φιλόδοξους για την πολιτική αυτή. Εγώ πιστεύω ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι ανάλογος των ε, φιλοδοξιών ακριβώς που έχουμε θέσει. Η διεύρυνση έλαβε χώρα με το ίδιο περίπου επίπεδο δαπανών για την κοινή αγροτική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Ζητάμε λοιπόν από τους γεωργούς να κάνουν περισσότερα και με την ίδια οικονομική απόδοση, ανάλογα με τον προπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα μπορούμε να περιμένουμε από την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή είναι η απάντησή μου στην ερώτησή σα. Ε, για ακριβέστερη απάντηση θα πρέπει να περιμένετε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Καθώ γνωρίζουμε ότι οι σημερινέ οικονομικέ συνθήκε είναι δυσχερεί. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τι δυνατότητε που μα προσφέρει ο προπολογισμό. Θα πρέπει με αποτελεσματικό τρόπο να διαχειριστούμε του πόρου του προπολογισμού στην γεωργία και για του παραδοσιακού κλασικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για του στόχου που έχουμε θέσει για το μέλλον με προοπτική το 2020. Θα πρέπει επίσης να πω και να τονίσω ότι Εάν υπάρξει μείωση των πόρων ε, τη κοινή αγροτική πολιτική, θα πρέπει να περιορίσουμε και τι φιλοδοξίε μα αναλόγω. Διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από του γεωργού να κάνουν περισσότερα, ούτε να του το ζητάμε αυτό, ε, με λιγότερη στήριξη. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, που είναι σκληρή. Του ζητάμε πολύ περισσότερα από ό,τι από του γεωργού στον υπόλοιπο κόσμο, με τέτοιου στόχου που έχουμε. Άρα θα πρέπει αναλόγω να προσαρμόσουμε, να είμαστε σαφεί και ξεκάθαροι. Εάν θέλουμε να έχουμε του ίδιου στόχου στην Ευρώπη, αλλά και να διατηρούμε του φυσικού πόρου ε, και να έχουμε βιώσιμη διαχείρισή του και να εργάζονται αποτελεσματικά οι γεωργοί, θα πρέπει να στηρίξουμε την γεωργία. Για την κοινοτικοποίηση λοιπόν τη κοινή αγροτική πολιτική, πρόκειται για μία από τι πιο εναρμονισμένε, τι πιο κοινοτικέ πολιτικέ που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη διάρθρωση που έχουμε σήμερα υπάρχουν δύο πυλώνε. Ένα πυλώνα που επικεντρώνεται στην ε, ε, αμοιβή των ε, δημοσίων υπηρεσιών και τη στήριξη που παρέχεται στου γεωργού. Σα θυμίζω εδώ ότι ο τομέα τη γεωργία είναι ο τομέα που έχει την ε, ύψιστη απόδοση, μάλλον κατά μέσο όρο απόδοση σε μείωση. Εδώ λοιπόν χρειάζεται απευθεία στήριξη και έχουμε και την απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών για τους γεωργού που δρούν στην ενιαία αγορά, που εκεί αναπτύσσουν τις δραστηριότητε τους. Ο πρώτος λοιπόν πυλώνα, ένα πυλώνα που 100% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έπειτα υπάρχει ο δεύτερο πυλώνα, ο οποίο ε, καλύπτει και τι εδαφικέ διαστάσει, τα ειδικά χαρακτηριστικά τη μια και τη άλλη περιοχή. Αυτό ο δεύτερο πυλώνα συγχρηματοδοτείται. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε συγχρηματοδότηση και στον πρώτο πυλώνα, θα πρέπει να δούμε αν από νομική άποψη μπορούμε να επιβάλλουμε στα κρατημέλη μελη συγχρηματοδότηση των εθνικών πολιτικών. Εάν δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν ή και όχι ανάλογα με του διαθέσιμου πόρου στον προπολογισμό του. Εδώ μπορούν να υπάρξουν αποκλήσει στο επίπεδο στήριξη των γεωργών που δρούν στην ενιαία αγορά. Και αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη και γι' αυτό ακριβώ πιστεύω ότι η διάρθρωση του πρώτου πυλώνα με 100% χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο και με δεύτερο πυλώνα συγχρηματοδοτούμενο εφόσον έχει να κάνει και με τους εδαφικού στόχους, νομίζω ότι αυτή η διάρθρωση είναι λειτουργική. Για το πώ έχει διαμορφωθεί ο προπολογισμό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τα μελετήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε τι διάφορε δυνατότητε και θα τα ε, παρουσιάσουμε με τη δημοσίευση τη ανακοίνωση για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Πάντω, σήμερα μπορώ να σα πω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η κοινή αγροτική πολιτική από τη μια είναι ε, ιστορικώ κοινοτική πολιτική, ε, ξεχωριστή, με στόχου που ορίζονται από την ίδια τη συνθήκη. Από την άλλη, όμω, ανταποκρίνεται και σε στόχου που έχουν ε, να κάνουν με τη στατική του 2020. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε ότι δεν γίνεται να την εξαρτήσουμε πλήρως από τη στατική του 2020. Υπάρχουν πολλά στοιχεία της κοινής αγροτικής πολιτικής που ε, εμπλέκονται με τη στρατηγική αυτή, αλλά όχι αποκλειστικώ. Ε, για την ε, συνοχή, την εδαφική συνοχή και την ύπεθρο. εδώ ήδη έχουμε συζητήσει με τον αρμόδιο επίτροπο στο επίπεδο του κολεγίου και πιστεύουμε ότι από αυτήν την έννοια θα πρέπει η ανάπτυξη τη υπαίθρου να μείνει ξεχωριστή από την εδαφική συνοχή με ξεχωριστό κανονισμό, με ξεχωριστό ταμείο και πόρου, με ξεχωριστού στόχου. Όμω θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο παραλληλισμό με κοινό κοινοτικό πλαίσιο που να επιτρέπει την επιδίωξη κοινών στόχων και περισσότερη συνέπεια στη χρήση των διαφορετικών μέσων, των διαφορετικών μέσων που προσφέρονται. Νομίζω ότι αυτή είναι η οδό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ακριβώς 10 λεπτά, πραγματικά 10 λεπτά μιλήσατε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν ε, θα λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι των ε, πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ, ο κύριος Αλπέρτ ε, Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και θα ήθελα να πω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, ε, κύριε Επίτροπε, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, θέματα όπου δεν αναφερθήκατε με λεπτομέρειες. Δηλαδή, για μας, εκείνο που ενδιαφέρει κυρίως είναι στο μέλλον. Ποιοι θα είναι οι πόροι εκείνοι που θα διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αγροτική πολιτική. Ακούμε διάφορες συζητήσεις. Ε, Μελικοί λένε 85%, άλλοι πάλι λένε 1%. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, κατά τη δική σας γνώμη, ποιο είναι το ποσοστό εκείνο το οποίο θα διατίθεται για την κοινωνική πολιτική στον προπολογισμό. Και μετά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Για ποιο ε, οικονομικό έτος μιλάμε. Άλλος μιλάει για πέντε, άλλος για επτά, άλλος ε, για δέκα χρόνια με ενδιάμεση εξέταση μετά από πέντε χρόνια. Αυτό είναι καθοριστική σημασία σε θέμα. Ε, γι' αυτό λοιπόν ρωτώ όσον αφορά την επόμενη οικονομική περίοδο Πώς ακριβώς μπορούμε να προγραμματίσουμε. Είπατε κι εσείς μόνο σας ότι αυξήθηκε ο αριθμός ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε και τα νέα κρατημέλη. Και εμείς ως ε, πολιτικοί για θέματα γεωργίας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στα 27 κρατημέλη ποικίλει κατά πολύ. Στη μεταρρύθμιση λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη τα οποία είναι στον πρώτο πυλώνα πολύ χαμηλά στις αποδόσεις ανακτάριο και στα υπόλοιπα. Εσείς λοιπόν τι είδους προγράμματα έχετε έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια ισορροπία στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, θίξατε το θέμα της ασφάλειας των ε, τροφίμων. Εγώ μόλις είχα κάποιες συζητήσεις από αυτού και θέλω να πω ότι στο μέλλον οφείλουμε να μεριμνήσουμε για 500 εκατομμύρια πολίτες να υπάρχει εξασφάλιση όχι μόνο της ποιότητας αλλά και της ποσότητας στον εφοδιασμό. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη ζάχαρη έχουν εξαντληθεί, έχουν πολιθεί όλες οι ποσότητες στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα της ζάχαρης είναι ένα θέμα. Και για σκεφτείτε πριν από έξι χρόνια συζητάγαμε για τη μεταρρύθμιση αγοράς στη ζάχαρη και τότε έγιναν παρατηρήσεις ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζαχαρότευτλων είναι πλέον περί τι, ότι δεν χρειάζεται πλέον τόση μεγάλη ποσότητα ζάχαρης ε, στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν <clears throat> πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε καλλιέργεια ζαχαρότεφλων και ζάχαρη στην Ευρώπη. Και επίση ε, πρέπει οι Ευρωπαίοι γεωργοί στο μέλλον, ε, όπω σα είπα, να μπορούν να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό για 500 εκατομμύρια κατοίκου. Εγώ ε, σα στηρίζω κύριε Επίτροπε και η δική μου πολιτική ομάδα θα σα στηρίξει, αλλά μην ξεχνάτε υπάρχουν πολλέ συζητήσει με αντικείμενο το ότι γιατί η κοινή αγροτική πολιτική καταλαμβάνει τόσο μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού στην Ευρώπη και απαντήσατε. Είπατε ότι η αγροτική πολιτική είναι ο μόνος τομέας που είναι σχεδόν απόλυτα κοινοτικοποιημένος. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κοινωνική πολιτική, την πολιτική παιδεία, έρευνα, στρατιωτικές δαπάνες. Υποτίθεται όλα αυτά θα ρυθμίζονται και από, από τις Βρυξέλλες. Κατόπιν τούτου το ποσοστό της κοινή γεωργικής πολιτικής θα είναι ελάχιστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές όμως ότι θα υπάρχει και μεγάλη κινητικοποίηση γιατί ε, κατά τη δεκαετία του 70 μιλάγαμε για ένα ποσοστό στον προπολογισμό της τάξης του 90%. Εμείς λοιπόν ως πολιτική ομάδα θα σας στηρίξουμε. Ε, θα τελειώσω κυρία Πρόεδρε, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Εγώ θέλω να κρατήσω το χρόνο μου. Κύριε Επίτροπε, εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε ένα σύστημα όπου μέσα στην Ευρώπη θα υπάρχει μέρημνα έτσι ώστε οι γεωργοί να αντιμετωπίζουν παντού παντού τις ίδιες προϋποθέσεις και συνθήκες. Να έχουμε μια ισορροπημένη ενιαία αγορά στα 27 κράτη-μέλη. Και μια ερώτηση κύριε Επίτροπε. Εσείς τι πιστεύετε αυτήν την αγορά στην Ευρώπη ε, μπορούμε κάπως να την προστατεύσουμε και σε σχέση με την ε, ταυτότητα και τη διατήρηση της ταυτότητας ε, των κρατών μελών. Υπάρχει κάτι που με απασχολεί και αυτό θα το δούμε και τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, ποια μέτρα μπορούμε εμείς ε, ως Ευρωπαίοι να λάβουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον ε, ε κατακλυσμό, την επίθεση των κερδοσκόπων στις πρώτες ύλε στη Γεωργία. Αυτά ήθελα να πω γιατί ήθελα να κρατήσω και το χρόνο που μου είχατε διαθέσει να μιλήσω. Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, Στέφαν Λεφόλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Πρώτα απ' όλα η τροφιμική ασφάλεια. Η ασφάλεια εφοδιασμού. Η κρίση που διατρέχουμε σήμερα καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε μια αγροτική πολιτική η οποία θα εξασφαλίσει την τροφιμική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και θα συμβάλλει στην ασφάλεια για όλο τον πλανήτη μας. Δεύτερο σημείο, <clears throat> όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος, υπάρχει το ζήτημα του περιβάλλοντος. Πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής και εξάλλου είναι τμήμα του εγχειρήματος Ευρώπη 2020. Είναι ο πρώτος μας στόχος. Τρίτος στόχος. Η, το σημείο, η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει μία συνιστόσα πολυμορφίας. Ορεινή γεωργία, γεωργία του κάμπου, γεωργία των ε, χορτολιμών, χορτολιβαδικών εκθράσεων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διατήρηση της πολυμορφίας, της γεωργίας και όλου του ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου. Αυτό είναι το τρίτο σημείο. Τέταρτο σημείο. Η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στις επιλογές της, συγκεκριμένα στην επιλογή να έχει μια γεωργική πολιτική και μια αγροτοτροφημική βιομηχανία που παράγει προϊόντα ποιότητος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κεφαλαιόδες για τη στρατηγική μας όταν θέλουμε να δούμε ποια πρέπει να έχουμε σε διεθνές επίπεδο για εμάς τους σοσιαλιστές αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα της κρίσης που έχουμε σήμερα που θέτουν και το θέμα της απασχόλησης. Και όπως είπε ο κύριος Επίτροπος, η γεωργία μαζί με την αγροτοτροφημική βιομηχανία είναι ο πρώτος εργοδότης στην Ευρώπη σήμερα και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Πέραν αυτού τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν, ποιες είναι, ποια τα συμπεράσματα στα οποία πρέπει να καταλήξουμε. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πρέπει να δεχτούμε οποιαδήποτε μορφή περικοπής του προπολογισμού της κοινή αγροτικής πολιτικής. Για οποιοδήποτε λόγο. Το τόνισε και ο κύριος Γκαρίγκα στην εισαγωγή του. Ορισμένοι θέλουν να μειώσουν τον προϋπολογισμό της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε πλήρω τον προπολογισμό όπω έχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θέλουμε οποιαδήποτε μείωση στον προπολογισμό τη γεωργίας. Δεύτερον, για του στόχου αυτού που και χρειαζόμαστε τον προπολογισμό έτσι κι αλλιώ για του στόχου μα. Δεύτερο θέμα είναι η συγχρηματοδότηση. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπερβούμε το τωρινό επίπεδο συγχρηματοδότηση γιατί αλλιώ θα μα φέρει αυτό σε μια διαδικασία επανεθνικοποίησης τη κοινή αγροτική πολιτική, κάτι το οποίο επέχει πάρα πολλού κινδύνου. απλού κινδύνους. Η Ευρώπη δηλαδή μπορεί να οδηγηθεί σε ένα ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών της. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ιδέα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και της συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γεωργία είναι τμήμα αυτού του εγχειρήματο. Πρέπει να υπερασπιστούμε μια κοινή αγροτική πολιτική σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση. Γι' αυτό δεν θέλουμε αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότηση. Τρίτο σημείο. Ήκοθεν νοείται ότι η ενσωμάτωση της γεωργίας στην οικονομία μας και στο παγκόσμιο επίπεδο προϋποθέτει κάποια στρατηγική και τη θέληση της Ευρώπης να παράγει, αλλά κυρίως να διατηρήσει το σήμα ποιότητας που έχει σε δυνατές επίπεδο. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Πρέπει σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπερασπιστούμε όλα αυτά τα στοιχεία που διατηρούν την ποιότητα και την ανεχνευσιμότητα των προϊόντων και η πρόσφατη κρίση με τη διοξίνη δείχνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επάγρυπνοι. Και επειδή τελειώνει ο χρόνο μου, θέλω να τονίσω επίση ότι πρέπει στα πλαίσια τη προστασία του περιβάλλοντο, στο στόχο αυτό του περιβάλλοντο, να έχουμε και την απαραίτητη φιλοδοξία για την πολιτική γεωργία, λαμβάνοντα υπόψη και τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη απλοποίηση των διαδικασιών. Υπάρχει σύγχυση σήμερα μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν και να πρασινίσουμε μέσα εισαγωγικά τον πρώτο πυλώνα και να διευκρινίσουμε καλύτερα τις αρμοδιότητες του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Ο πρώτος δηλαδή να έχει όλες τις αιτήσιε επιδοτήσει και ο δεύτερο να έχει επιδοτήσει οι οποίε έχουν συμβατικό χαρακτήρα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να χαράξουμε τις πολιτικές μας, τις κατευθύνσεις για την κοινή αγροτική πολιτική και τα συμπεράσματα που πρέπει να προκύψουν στο επίπεδο του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις οικονομικές διαστάσεις ε, της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η Επιτροπή μας παρουσίασε πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα κατά τους τελευταίους έξι μήνες και είναι ενδιαφέροντα κάτω από το πρίσμα της γεωργικής πολιτικής. Βεβαίως λείπουν κάποια στοιχεία που αφορούν ε, στην, ε, στην γεωργική μεταρρυθμίση. Ε, υπάρχουν συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, διαβουλεύσεις για τον προπλογισμό του 2011 που δείχνουν ότι ανησυχούμε πάρα πολύ κρατημέλη για τις δαπάνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 18 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ε, λάβαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή. Η επιστολή μάλιστα απευθυνόταν προς την Επιτροπή όπου οι πρωθυπουργοί μεταξύ αυτών της Γαλλίας, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της δικής μου της χώρας, της Φινλανδίας, όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί ε, ζητούν ε, να υπάρχει μια προσαρμογή στον προϋπολογισμό. Ε, ζητούν ε, εκτόσεις ε, γεωργικές μεταρρυθμίσεις. Εκεί στην επιστολή μπορείτε να διαβάσετε και τις απόψεις της δικής μου της κυβέρνησης. Γνωρίζοντας όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ δεν χαίρομαι, δεν μ' αρέσει αυτό κράτη-μέλη να γράφουν επιστολές στην Επιτροπή για να τις δίνουν καλές συμβουλές και δεν νομίζω ότι αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα και την Κομισιόν. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στην Επιτροπή ε, όπου προετοιμάζεται η γεωργική μεταρρύθμιση θα πρέπει να λάβουν χώρα ε, και να ληφθούν υπόψη κάποιες ισορροπίες. Το ΙΛΚ αναφέρθηκε στο ότι οι άμεσες ε, καταβολές θα πρέπει να είναι πιο δίκαιες, τουλάχιστον όσον αφορά τα νέα κράτη-μέλη. Ε, αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της ε, πολιτικής που εφαρμόζεται ίσως πράγματι να μην υπάρχει κάποια ισορροπία. Επειδή λοιπόν εστάλει αυτή η επιστολή και επειδή υπάρχει και αυτό που σας είπα ε, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τους πόρους για την κοινή γεωργική πολιτική. Θα μας ενδιαφέρει η Κομισιόν να σχολιάσει όλα αυτά. Οι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι είναι επίση απαραίτητο να υπάρξουν και συγκεκριμένες περικοπές μέσα στην κοινή γεωργική πολιτική να έχουμε μια πιο δίκαιη πολιτική γιατί δεν μπορούμε ε, να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε περισσότερους πόρους στο μέλλον από αυτούς που έχουμε τώρα. Και δυστυχώς μερικές φορές φοβάμαι, εξακολουθεί να υπάρχουν κάποιοι, ότι ε, θα ισχύσουν το να έχουμε περισσότερους πόρους. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Η κοινή πολιτική δεν μπορεί να διωγγωθεί περαιτέρω. Υπάρχουν μάλιστα πιέσεις η πολιτική να ακολουθήσει την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και επειδή υπάρχουν όλα αυτά θα ήθελα ο Επιτρόπος να σχολιάσει. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα με ενδιέφερε να γνωρίζω ε, κατά πόσο η πολιτική ε, θέλει να σχολιάσει ε, την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει την πολιτική για το 2020. Μέχρι τώρα έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα ότι είναι σημαντική η πολιτική αυτή, αλλά θα ήθελα να υπάρξουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα μας ενδιέφεραν όλα αυτά εκ μέρους των φιλελευθέρων. Vielen Dank. Jetzt Bas für die Grünen. Η πράσινη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, παρουσίασή σας. Για εμάς του πρασίνου υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συμφωνώ μαζί σας κύριε Επίτροπε. Ναι, χρειαζόμαστε μια αλλαγή στι τωρινέ αγροτικές πολιτικές. Ζητάμε κάτι περισσότερο από τους αγρότες μας στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν παράλληλα περικοπές αν θέλουμε να παράχουν, να περαιτέρω υπηρεσίες, πρέπει να έχουν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αυτό είναι σημαντικό σημείο αναφοράς. Αλλά αν θέλουμε να ενισχύσουμε την αγροτική πολιτική πρέπει κάτι να αλλάξει. Η πρώτη επιλογή σας μεταξύ αυτών που αναφέρατε τον Νοέμβριο, η πρώτη επιλογή, το business as usual, αυτό δεν είναι πραγματική επιλογή. Ξέρουμε όλοι ότι οι επικρίσεις για τις τωρινές πτυχές της πολιτικής γεωργίας είναι πολύ σημαντικές, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως είπε και ο Καρλ, αν υπάρξει μεγάλη πίεση στον προϋπορισμό όπως σήμερα, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε με τα δημόσια χρήματα τα οποία οδηγούν σε δημόσια αγαθά. Αυτό θα πρέπει να είναι η κύρια γραμμή τη αγροτική μα πολιτική. Το business as usual, λοιπόν, η συνέχιση τη τωρινή κατάσταση δεν είναι επιλογή για του πράσινου οι άλλες δύο τώρα επιλογές που αναφέρατε στην ανακοίνωσή σας, εκεί υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε. Στη δεύτερη παραγωγή χάρη μιλάτε για πρασίνισμα των αμέσων πληρωμών. Τι σημαίνει όμως αυτό. Δεν είναι σαφές. Για μας τους πρασίνους θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο την, ποιότητα των, την ποσότητα των γεωργικών προϊόντων αλλά και την ποιότητά τους και αυτό είναι κομμάτι της στρατηγικής του 2020 και αυτό σημαίνει πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων. Εδώ η γεωργία παίζει ένα σημαντικό ρόλο ο οποίο είναι κομβικό αν μιλάμε για το πρασίνισμα των πρασίνων των ε, αμέσων πληρωμών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά. Περνόμαστε πιο συγκεκριμένοι στο τι σημαίνει το πρασίνισμα των άμεσων πληρωμών. Τέλος, μιλήσατε και για τους γεωργού και τις επιδοτήσει για του μικρούς γεωργού. Αλλά όταν σας ρωτάμε τι ακριβώς εννοείτε, λέτε εξυγχρονισμό των μικρών γεωργών. Τι θα πει αυτό. Σημαίνει την βιομηχανοποίηση της γεωργίας που βλέπουμε σε χώρες όπως η δική μου, οι κατοχώρες. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αν αυτό σημαίνει ότι οι μικρογεωργοί θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κλιματική αλλαγή και να έχουν καλύτερη χρήση πόρων, τότε ναι, αυτό είναι πραγματική υποστήριξη για τη διατήρηση των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα είναι σε καλύτερη θέση να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό το υποστηρίζουμε. Δεν υποστηρίζουμε απλώ όμω μια περαιτέρω βιομηχανοποίηση των μικρών γεωργών. Αυτό δεν είναι εξυγχρονισμό για μα. Αυτό είναι επιστροφή στο παρελθόν. Επίσης ένα σημαντικό θέμα για μας είναι η γεωργή σε μειονεκτικές περιοχές που είναι σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι επιδοτήσεις για αυτούς τους γεωργούς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτά για τον πρώτο πυλώνα λοιπόν. Δεύτερος πυλώνας. Μιλάμε για την αγροτική ανάπτυξη εδώ. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να συνδέεται πολύ περισσότερο με την περιφερειακή ανάπτυξη. Εσείς είπατε, χρειάζεται περισσότερο συντονισμός μεταξύ του Ταμείου Συνοχής και του Αγροτικού Ταμείου. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα όραμα για την εδαφική συνοχή να μιλάει για δημόσια αγαθά τα οποία πρέπει να δίδονται στις περιφέρειες και εκεί μπορούμε να δούμε πώς θα πρέπει να συμβάλλει το Αγροτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Αν το δούμε αυτό λοιπόν υπό την οπτική γωνία της εδαφικής συνοχής, συμφωνώ μαζί σας. Μία επίκριση τώρα δεν αναφερθήκατε καθόλου σε ό,τι αφορά την επίπτωση της κοινή αγροτικής πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πράσινους. Για μας ένα από τα κέρια θέματα για την ΚΑΠ είναι το ότι ο αντίκτυπος των πολιτικών μας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οποιαδήποτε μορφή dumping αγροτικών προϊόντων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να σταματήσει, να εγκαταληφθούν οι επιδοτήσει εξαγωγή. Εμεί επηρεάσουμε αρνητικά τι οικονομίε του, και αυτό σίγουρα δεν είναι θετικό, είναι μια αντιμετώπιση 19ου, 20ου άντε αιώνα, αλλά όχι 21ου αιώνα. Αυτό σημαίνει πρέπει να βοηθήσουμε γεωργού γεωργούς αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν και περισσότερη προστιθέμενη αξία και όχι μονάχα να στέλνουν εδώ μονάχα τα βασικά του προϊόντα και εμεί να καρπούμεθα την προστιθέμενη αξία. Όχι, θα πρέπει η προστιθέμενη αξία να καταλήγει σε αυτέ τι χώρε. Είμαι ακριβώς εκεί που θέλετε να φτάσετε σχεδόν. Χαίρομαι που σας ενδιαφέρουν αυτά που λέω. <clears throat> Τελευταίο σημείο. Είναι περίπου και το σημείο κίνησης. Αν ζητάμε περισσότερα από τους γεωργούς θα πρέπει να δούμε ποια είναι και η θέση των γεωργών. θα πρέπει να είμαστε σε θέση να του βοηθήσουμε να αναπτυχθούν καλύτερα σε οργανώσεις παραγωγών και να δούμε και ποια είναι η θέση του λιανικού εμπορίου σήμερα στα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει πάντα μια πίεση κατά των γεωργών από τα σούπερ μάρκετ και τους λιανοπολιτές. Ζητάμε πάρα πολλά από αυτού και αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανωθούν λίγο καλύτερα σε οργανώσεις παραγωγών για να έχουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση και να διατηρήσουν μια ισχυρή και αηφόρο γεωργία. Και το αφήνω στο συναδελφό μου να συνεχίσει. für die ECR. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρέμβαση μιλώντα εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, να πω ότι για μα είναι προφανές, στην ομάδα μας, ότι το συνολικό μέγεθος του, του ευρωπαϊκού προπολογισμού εντός του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα παγώσει. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό με τον προπολογισμό, προκύπτει και το εξή προφανές... Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική που καλύπτει το 42% των σημερινών δαπανών θα αντιμετωπίσει μεγάλο ανταγωνισμό από άλλες ε, από άλλου τομεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτούν και εκείνη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθεί σε κρίση. Υπάρχουν 23 εκατομμύρια άνθρωποι που θα βρεθούν εκτό ε, αγορά εργασία. Εδώ όμω θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότητα. Είναι λοιπόν ε, ορθόν ότι θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασχοληθεί με όλες αυτές τις προκλήσεις. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που μας δίνει η στρατηγική της ε, του 2020. Το καλό, η καλή είδηση για την κοινή αγροτική πολιτική είναι ότι έχει σημαντικό ρόλο να διδραματίσει εντό τη στρατηγική του 2020. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί εντό ενό εξελισσόμενου κόσμου, με έναν πληθυσμό που ολοένα αυξάνεται και είναι και πιο εύκολο, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων. Η επισητιστική ασφάλεια θα γίνει ένα τεράστιο θέμα μέχρι το τέλο αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου. Άρα η παραγωγή τροφίμων και η γεωργική παραγωγή θα είναι στρατηγική σημασία και ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα η γεωργία και η ανάπτυξη τη υπαίθρου θα πρέπει να προσφέρουν κοινά ωφέλη, δημόσια ωφέλη στους πολίτες όπως ορθώ τα αναμένουν. Και εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι προκλήσει των κλιματικών αλλαγών. Τώρα επειδή η γεωργία και η ανάπτυξη τη υπαίθρου συμβάλλουν ε, μέγιστα στην ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να διασφαλίσουμε τι θέσει εργασία που δημιουργούνται στην Ήπεθρο και στον χώρο τη Γεωργία. Η κακή είδηση βέβαια είναι ότι εδώ απειλούνται όλα τα επιτέχματα της ευρωπαϊκής γεωργίας του παρελθόντος. Διότι η ευρωπαϊκή Δημηχανία γεωργική Δημηχανία δεν αυξάνεται με, αρκετά γοργούς ρυθμούς. Ε, το μέσο εισόδημα του μέσου γεωργού ε, σήμερα είναι 15% λιγότερο από τον μέσο ευρωπαίο εργαζόμενο. Άρα η ευρωπαϊκή γεωργική βιομηχανία απέχει πολύ από το να είναι μια αυτάρκης, να είναι ένας αυτάρκης και αυτοχρηματοδοτούμενος ε, βιομηχανικός κλάδος. Χρειάζονται ακόμη εδώ στήριξη και επιδοτήσεις. Και είναι μια βιομηχανία με μεγάλο κόστος. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευάλωτη στον διεθνή ανταγωνισμό. Ε, και ο ανταγωνισμός αυτός δεν θα πάψει να αυξάνεται καθώς απελευθερώνεται όλο και περισσότερο το διεθνές εμπόριο. Εν τω μεταξύ, για τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ του υψηλού επίπεδου ε, ε, των υψηλών επίπεδων βοηθειών που δίνονται σε κάποιους ε, κλάδους. Ε, στα παραδοσιακα κάτι κράτη-μέλη και τις άλλες βοήθειες που δίνονται σε νέα κράτη-μέλη με τομεί που δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί και συχνά δημιουργούν προβλήματα. Αυτά θα μπορεί να ληφθούν υπόψη στη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική, λαμβάνοντα υπόψη τη μεγαλύτερη ζήτηση με τον συρρυκνούμενο προπολογισμό. Επιμένω λοιπόν, Πρόεδρε, ότι εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την ε, ανάγκη να στηρίξουμε την κοινή αγροτική πολιτική. Και εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα. Ε, κοινή αγροτική πολιτική και ο κόσμο τη Πέτρου θα παραμένουν ένα ε, βαρύνων κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όμω, σε όλη τη διάρκεια αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των δαπανών, την προστιθέμενη αξία και κυρίω του αν έχουμε όφελο για τα χρήματα που δαπανούμε έχουμε εξετάσει κάποιε τέτοιε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προτινόμενη μεταρρύθμιση και εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει επαρκέ όραμα και ικανοποιητική στόχη για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Γεωργική Βιομηχανία. Δεν καλύπτουν τι προσδοκίε των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα αυτό, δεν καλύπτουν του στόχου αύξηση τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Γεωργική Βιομηχανία και σε αυτού του απαιτητικού ε, καιρού θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όχι μόνο χρειάζεται όραμα και φιλοδοξίε για τη μεταρρυθμιζόμενη αυτή η γεωργική βιομηχανία, θα πρέπει να αποδείξει και στο κοινό, στου πολίτε, ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκή αγροτικής Βιομηχανία θα δώσει αξία για τα χρήματα που δαπανώνται, όχι μόνο ε, ότι θα παραμείνουμε στην προσφορά κονδυλίων. Αν κοιτάξω γύρω μου, βλέπω ότι δεν υπάρχει κανείς από την ΚΟΥ εδώ, ο οποίος «Α, είσαστε εδώ, βεβαίως». Βρήκαμε κάποιον από την ΚΟΥΕ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας είπα προηγουμένως, μάλλον είπα στη γραμματεία ότι θα μιλήσω εγώ εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, αλλά ίσως η γραμματεία δεν το κατάλαβε. Εξ ονόματος λοιπόν της Ενωμένης Αριστεράς θέλω και εγώ να δώσω μια απάντηση στα εισαγωγικά σχόλια της Κομισιόν. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τον κύριο Επίτροπο. Θέλω να πω όμως ότι για μας το βασικό στοιχείο της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι η αλληλεγγύη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η γεωργία δεν είναι μονάχα μια απλή αγορά. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πρέπει να υπάρξει αρρωγή προς τους γεωργούς με τον ένα τρόπο με τον άλλο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης και την, τις διαφορές, τις ανισότητες που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Έκεν. Επίσης η αλληλεγγύη πρέπει να στρέφεται και προς τα έξω και προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν πρέπει η κοινή αγροτική πολιτική να μα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου θα κάνουμε πρακτικές dumping των αγροτικών μας προϊόντων μέσω των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Και έτσι αναχαιτίζουμε και αναστέλουμε την οικονομική ανάπτυξη στις ε, χώρες αυτές σε ό,τι αφορά το γεωργικό τομέα. Επίσης φαίνεται να υπάρχει σύγχυση σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινή αγροτική πολιτική. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο συντηρητικό μου συνάδελφος, <clears throat> λέγοντας ότι δεν είναι πολύ σαφές από την ανακοίνωση της Κομισιόν προ τα που θέλει η Κομισιόν να κινηθεί. Πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Έχουμε τις ε, τέσσερις κατευθύνσεις χρηματοδότησης κοινής αγροτικής πολιτικής, ε, εξισορρόψης αγοράς, άμεσες επιδοτήσεις προς τους ε, γεωργούς που φυσικά έχουν και το χαρακτήρα της αλληλεγγύης κυρίως είναι το γεωργό στις χώρες που η γεωργία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη και ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι η προστασία του περιβάλλοντος και το τέταρτο σημείο το οποίο αναφέρθηκε και είναι εξίσου σημαντικό είναι ανάγκη να προχωρήσουμε και σε καινοτομία στον τομέα της γεωργίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά και είναι αλληλένδετο με την αποτελεσματικότητα του αγροτοτροφημικού τομέα στην Ευρώπη του μέλλοντος. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την ΚΑΠΑ, αλλά είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να πράξει η ΚΑΠΑ επομένως. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους πολιετής μας προϋπολογισμούς και καλύτερη στοχοθεσία. Και από τη μία μεριά αυτό συνεπάγεται την ε, διασύνδεση με το Ταμείο Συνοχής και τους στόχους της αλληλεγγύης. Πολύ περισσότεροι γεωργοί πρέπει να έχουν υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε όχι μόνο μικρούς γεωργούς στην Ευρώπη, αλλά και τεράστιες αγροτοτροφημικές επιχειρήσεις. Και φαίνεται ότι ο ενδιάμεσος χώρος αρχίζει πια να εξαφανίζεται ή έχουμε μικρούς γεωργούς ή μεγάλες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της συνοχής θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους μικρούς γεωργούς, ιδίως στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται ακόμα να υπάρξουν διορθωτικές ενέργειες στη λειτουργία της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Και η καινοτομία είναι σημαντικός στόχος. Θα πρέπει να δούμε τι χρηματοδότηση υπάρχει για τη βελτίωση της καινοτομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως μέσα στα πλαίσια τη γεωργίας και όχι να έχουμε αυτόνομη χρηματοδότηση τη καινοτομία στον ε, τομέα της ΚΑΠ. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στον τομέα της γεωργίας και για την αηφορία. Οι μικρές επιχειρήσεις ιδίω θα πρέπει να διατηρηθούν γιατί πρέπει να διατηρηθεί ο σημαντικός τους ρόλος στην διαχείριση της αγροτικής πολιτικής. Θα πρέπει να αμυφθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν αυτές οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και στο περιβάλλον, στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Όταν βλέπετε τι χαρτοβασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει ένα μικρό γεωργό στην Ευρώπη, αυτό δεν είναι αποτελεσματικό και καθόλου λυσιτελέ. Δεν μα οδηγεί σε μία επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον που είχαμε θεσπίσει εμεί. οι δεν σημαίνει ότι τα κάτι μέλη θα πρέπει να βρίσκουν εδώ και εκεί περιοχές ε, χρηματοδότησης. Αλλά σίγουρα πρέπει οι γεωργοί να εξασφαλίσουν την υπηρεσία προς το περιβάλλον και να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι εμείς δεν στηρίζουμε την ΚΑΠ, αυτό βέβαια το γνωρίζουν όλοι. Εγώ θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι ο πρόεδρος Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, επανειλημμένα έχει αναφερθεί στην προστιθέμενη αξία, στην επικουρικότητα και στην αλληλεγγύη. Θα ήθελα λοιπόν ο Επίτροπος να αναφερθεί στην προστιθέμενη αξία που προσέφερε η κοινή πολιτική τα τελευταία δέκα χρόνια. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια πολιτική, τότε πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης επιτυχημένο στο παρελθόν. Δεν είμαι λοιπόν καθόλου σίγουρη για το ότι σε αυτήν εδώ τη συζήτηση που γίνεται έχει λάβει η χώρα και μια ενδελεχής μελέτη ε, για το τι κρίθηκε επιτυχές τα τελευταία χρόνια, 10-20 χρόνια. Όσον αφορά την επιστολή των πέντε πρωθυπουργών και ε, αυτή η επιστολή συζητήθηκε, τέθηκα διάρκεια της συζήτησης και ρωτώ τον Επίτροπο τι είδους ε, μέτρα και αλλαγές προτίθεται να προτείνει για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με λιγότερους πόρους και τέλος ποια είναι η άποψη του Επιτρόπου ε, σχετικά με τον κατάλογο των αποδεκτών ε, που δημοσιεύτηκε εκεί φαίνεται είναι πρόδειλο ότι κάποιοι εξ αυτών δεν χρειάζονταν αυτή τη βοήθεια που τους χορηγήθηκε. Τώρα, ε, κλείσαμε με τις πολιτικές ομάδες και τώρα θα μιλήσουμε με τον, ε, θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής. Ευχαριστώ την πρόεδρο που μου δίνει την ευκαιρία να πάρω το λόγο σήμερα, να χαιρετήσω τον Επιτροπό και θα είμαι σύντομος, διότι ήδη εκφράστηκαν διασμοί και νομίζω με τρόπο πολύ ξεκάθαρο. Με την παρέμβαση μου θέλω να τονίσω το γεγονός ότι σήμερα μας απασχολούν τα κονδύλια. Τα κονδύλια θα πρέπει να αποδώσουμε στην κοινή αγροτική πολιτική και αυτό θα πρέπει να το δούμε από μια οπτική γωνία τελείως διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, μάλλον η εξέλιξη της κοινής αγροτικής πολιτικής τα τελευταία 20 χρόνια, ε, επηρεάζονται από τις ε, προτάσεις που έχουν γίνει για τη μεταρρύθμιση με σκοπό να οικοδομηθεί μια πολιτική που να ξεφύγει από το στενό κύκλο των κοινοτικών πολιτικών και να καλύψει στόχους και φιλοδοξίες που θα εξυπηρετούν το σύνολο της, Ευρωπαϊκής, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ε, στόχους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, που των οποίων οι γεωργοί να γίνουν οι φυσικοί ερμηνευτές. Η διασύνδεση της γεωργίας με την εξοικονόμηση των υδάτων, τα εδάφη, τη βιοπικιλότητα, την προστασία των φυσικών πόρων είναι δημόσια αγαθά όλα αυτά που θα πρέπει να επιδιωχθούν σήμερα για την βιώσιμη και την ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας μας αξίες αυτές πρέπει να υποστηριχθούν και με πολιτικές και με πόρους κατάλληλους. Ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν από το 1992 οδήγησε σε σταδιακή μείωση των ε, πόρων που αποδίδονται ως τώρα στην πολιτική αυτή. Μια μείωση όλο και περισσότερο σημαντική εάν τη δούμε υπό το φως της ε, πορείας της διεύρυνσης με την έναρξη του νέου προγραμματισμού θα καταλήξουμε σε 29 πλέον κρατημέλη θα πρέπει λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις, χωρίς να έχουμε όμως άλλες περικοπές των πόρων της Γεωργίας. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου ε, τονίζει και έπειτα με μεγάλη πλειοψηφία γκρίναμε και την ε, πορεία αυτή μέσω της ε, έκθεσης του συναδέλφου Λάιον. Και βεβαίω το Μάρτιο ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε και την ανάλογη έκθεση του συναδέλφου Ντε. Τον περασμένο Ιούλιο ε, εγκρίναμε ένα ενιολογικό πλαίσιο που ξεπερνά τελείω ε, την θεώρηση αυτή τη πολιτική που είχε να κάνει με την απλή στήριξη των γεωργών στην δραστηριότητά του. Σήμερα και η νέα αγροτική πολιτική εκπροσωπεί πολύ περισσότερα. Χρειάζεται μια εξαιρετική ε, έμφαση στο να δούμε τι προσδοκίε των πολιτών μα και των γεωργών, να καταλάβουμε καλύτερα του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη ευφυού ανάπτυξη που έχουμε θέσει ω πυρήνα τη στρατηγική το 2020. Εδώ θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την ιστορικώ σημαντικότερη πολιτική και λόγω τη ιστορία τη και λόγω του κύρου και του βάρου τη. Ε, μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερη, διότι αυτή τη στιγμή η επιστημιστική ασφάλεια μα ε, απασχολεί ιδιαιτέρω, με ιδιαίτερη ένταση και κυρίω ε, σε σχέση με το μέλλον. Τι τελευταίε ημέρε είχαμε διαμαρτυρίε στην Αλγερία και την, ε, Ισία. Αυτέ είναι οι πρώτε εκδηλώσει ε, του γεγονότο ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Τα τρόφιμα κινδυνεύουν να γίνουν ένα αγαθό που θα μα λείπει. Στην Ευρώπη λοιπόν δεν μπορούμε να μελήσουμε την ανάγκη να δώσουμε μια στρατηγική απόκριση ε, και καινούργια απόκριση σε αυτήν τη νέα δυσκολία. Θα πρέπει τους πολίτες να τους απαλλάξουμε από αυτήν την επιπλέον δυσκολία, να τους διασφαλίσουμε. Και δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια, ένα σωστό πλαίσιο την κοινή αγροτική πολιτική και να ικανοποιήσουμε τι προσδοκίε των πολιτών έτσι όπω έχουμε ξεκινήσει χωρίς Ευρω... ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρί να ακολουθήσουμε του στόχου αυτού. Έχουμε 14 εκατομμύρια Ευρωπαίου Γεωργού σήμερα, τον οποίο πρέπει να σεβαστούμε τι απαιτήσει. Αυτοί σήμερα διαχειρίζονται το ίμιση τη επικράτεια τη Ένωσή μα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την απειλή, να μειωθεί ο ρόλο τη Ευρώπη, να καλύψουμε την φιλοδοξία να δημιουργηθεί μια Ευρώπη ισχυρή με περισσότερε αρμοδιότητε. Αυτέ οι μεγαλύτερε αρμοδιότητε δεν μπορούν να περνούν να μην λάβουν υπόψη μάλλον τον ε, ε, αυξανόμενο ανταγωνισμό για τους δημοσιονομικούς πόρους. Θα πρέπει απαραίτητο να αποδώσουμε μεγαλύτερους πόρους στην πολιτική αυτή και να ε, ακολουθήσουμε τις ανάγκες των δημοσιονομικών γραμμών. Θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να λάβουμε υπόψη αυτή την προοπτική και σήμερα με μια διαρθρωμένη συζήτηση να σκεφτούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλέψουμε μια ανταπόκριση στο ύψος των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Ja, vielen Dank. Ε, Merci, λέει η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει τελειώσει ο πρώτος Κύριε Επίτροπε, έχετε φυσικά τώρα την ευκαιρία να προβείτε σε μια πρώτη σειρά απαντήσεων και στη συνέχεια αρχίζει ο κατάλογος των υπολείπων ομιλητών. Είναι μακρύς ο κατάλογος 14 ονόματα έχω εδώ. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο και οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια θα είναι σύντομοι και συνοπτικοί και θα δώσουμε στη συνέχεια στον κύριο Επίτροπο τη δυνατότητα να απαντήσει και πάλι στο δεύτερο γύρο. Πρώτα όμως κύριε Σόλος έχετε το, το λόγο για τις πρώτες σας απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι ως δυνατόν πιο λακωνικός όσο είναι δυνατόν. Πρώτο ερώτημα, υποστήριξη της κοινή αγροτικής πολιτικής και αποδοτικότητά της τα τελευταία χρόνια. Σκεφτείτε ποιο θα ήταν το κόστος για την ευρωπαϊκή κοινωνία χωρίς την ΚΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τροφοδοσίας της αγοράς με τροφιμικά προϊόντα και επίσης υπό την έποψη της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Είναι εύκολο να το σκεφτόμαστε αυτό όταν υπάρχει η τροφιμική επάρκεια γιατί λειτουργεί η κοινή αγροτική πολιτική. Κοιτάξτε όμως τα μέσα ενημέρωσης τι λένε για τις περιοχές που δεν υπάρχει μια τέτοια πολιτική ή έχει άλλες κατευθύνσεις ποια είναι τα αποτελέσματα. Εγώ δεν θα ήθελα η Ευρώπη να βρεθεί σε αυτή την εμπειρία. Να μην έχουμε υποστήριξη στη γεωργία και να αναγκαστούμε να θέσουμε αυτό το ερώτημα σε κατάσταση κρίσης. Επομένως η Ευρώπη δεν αντιμετώπισε ποτέ προβλήματα τροφίμων τα τελευταία 50 χρόνια. Έχει τροποποιήσει πολλές φορές την κοινή αγροτική πολιτική για να την προσαρμόσει στις ανάγκες της αγοράς. Αν στη δεκαετία του 60 θέλαμε απλώς να έχουμε τρόφιμα. Στη συνέχεια υπήρξε και τροποποίηση αυτή τη ε, πολιτικής ότι ως είπε ο κύριος ε, πρόεδρος Δεκάστρο να προσαρμοστεί στην ανάγκη παραγωγή δημοσίων αγαθών. Ξέρουμε ότι οι γεωργοί πρέπει να μείνουν στην Ήπεθρο για να διατηρήσουν και το περιβάλλον και την αγροτική υποδομή η οποία χρειάζεται για την παραγωγή. Ο γεωργός <coughs> δεν παράγει γεωργικά προϊόντα από το πρωί στο μεσημέρι και το απόγευμα δημόσια αγαθά, άλλου είδους. Όλα αυτά είναι ολοκληρωμένα και ενσωματωμένα. Θα πρέπει να σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει κοινή αγροτική αγροτική πολιτική χωρίς κοινή αγροτική πολιτική. Σημαίνει συγκέντρωση αγροτικής δραστηριότητας μόνο στα έφορα εδάφη και στις παράκτιες περιοχές και συνολική εγκατάλειψη της γης σε όλα τα άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτό όμω θα σήμαινε απερίμωση του αγροτικού χώρου σε πολλά μέρη της Ευρώπης, γιατί χωρίς την αγροτική πολιτική και την αγροτική παραγωγή δεν θα υπήρχε παραμονή του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές αυτό θα σήμαινε επίσης και τεράστια πίεση στους φυσικούς πόρους, αύξηση της ρήπανσης, μείωση της γονιμότητας των εδαφών, βιομηχανοποίηση της γεωργίας. Εν καιρό λοιπόν θα είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα και για την ε, τροφοδοσία με προϊόντα ασφαλή και προϊόντα ποιότητος σε επαρκείς ποσότητες. <clears throat> Αυτή είναι λοιπόν η ενσυντομή απάντησή μου στο ερώτημα αυτό που τέθηκε. Πιο συγκεκριμένα ερωτήματα τέθηκαν επίση για το ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό τη κοινή αγροτική πολιτική στου μελλοντικού προπολογισμού. Ξέρουμε ποιο θα είναι το συνολικό ύψο των προπολογισμών. Είναι πολύ δύσκολο να, να μιλήσουμε για ποσοστά. Ένα πράγμα θέλω να υπογραμμίσω. Το να μειωθεί ο κοινοτικό προπολογισμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του προπολογισμού γεωργία. Σημαίνει απλώ μεταφορά στου προπολογισμού των κρατών μελών. Γιατί για πολλούς λόγους, εισόδημα των γεωργών, ισορροπία σε χωροταξικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που θέλουν να διατηρήσουν και να υποστηρίξουν τη γεωργία. Αναφέρθηκε το ποσοστό 39% του προϋπολογισμού, αλλά συγχρόνως λιγότερο από 1% στον, στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία. Αν μειώσουμε το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει αυτό μεγαλύτερη πίεση στου εθνικούς προπολογισμού αλλά και μείωση των κοινοτικών πολιτικών. Δεν μπορώ να σα πω λοιπόν ποιο θα πρέπει να είναι το επίπεδο του προπολογισμού. Σα λέω ποιε είναι οι φιλοδοξίε μα για τη μελλοντική πολιτική. <clears throat> αν, αν μειωθούν λοιπόν οι πόροι θα μειωθούν και οι ε, φιλοδοξίες μας και επομένως θα πρέπει να θεσπίσουμε κριτήρια τα οποία να εφαρμόζονται οριζόντια σε όλα τα κράτη-μέλη. Να σταματήσουμε να βασιζόμαστε μονάχα στην ιστορική βάση των επιδοτήσεων και όλα αυτά περιλαμβάνονται στις προτάσεις που θα διατυπώσει η Κομισιόν. Η απαραίτητη αυτή ισορροπία θα εξαρτηθεί τελικά από το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με το θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής και των δια διεθνών αγορών και τις κερδοσκοπίες της πρώτες ύλες. Αυτό δεν είναι μονάχα θέμα κοινή αγροτική πολιτική, είναι ένα θέμα συνολικό το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι G20 επίσης, οι οποίες συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη, θα πρέπει και αυτοί να προτείνουν λύσεις σε αυτό το παγκοσμίο πρόβλημα. Δεν επαρέχομαι στο θέμα της αποτυχίας της μεταρρύθμισης κοινή αγροτικής πολιτικής που ανεφέρθη από ορισμένου. Δεν ξέρω αν το γεγονό ότι έχουμε μια συνεχή τροφοδοσία των αγορών αποτελεί αποτυχία. Μπορούμε να μιλήσουμε για ανάγκη τροποποιήσεων και προσαρμογών που θα χρειαστούν και στο μέλλον όπως έγινε και στο παρελθόν. Πάντα υπάρχουν πράγματα να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν. Τίθεται το θέμα της καλύτερης κατανομής των κονδυλίων μεταξύ μικρών και μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων και το θέμα της ισοδικίας επιδοτήσεων μεταξύ νέων και παλαιών χωρών για να μην υπάρξει γεωργία δύο κατευθύνσεων και επίσης η καλύτερη κατεύθυνση της χρηματοδότησης ώστε να παράσχει κίνητρα για την καινοτομία μεταξύ των γεωργών για τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Όλα αυτά είναι αδυστήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω όμως ότι χωρούν λόγοι να μιλήσουμε για αποτυχία της κοινή αγροτικής πολιτικής όπως εξήγησα. Η σχέση με τη στρατηγική 2020, Ευρώπη 2020, όπως σας είπα, νομίζω ότι είναι σαφές ότι η γεωργική πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίσει την αηφόρο ανάπτυξη. Μιλάμε και για τον αγροτοτροφημικό τομέα που θα πρέπει να υποστηρίξει και την ε, καινοτομία χάρη στις επενδύσεις στον τομέα αυτό ο στόχο μας θα πρέπει να είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα <clears throat> του σύνολου αυτού τομέα με μια καλύτερη και πιο αηφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Η αηφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κοινή αγροτική πολιτική για του λόγου που σας ανέφερα προηγουμένω, γιατί όλη η γεωργία αλλιώ θα πήγαινε στα πιο έφορα εδάφη με τεράστια πίεση στου φυσικού πόρου. Στον αγροτικό τομέα επίση στον αγροτικό χώρο. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική που να εξασφαλίσει τη διατήρηση της, του πληθυσμού και του εισοδήματος των γεωργών στην περιοχή αυτή. Στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό είναι ήδη ενσωματωμένη σε μεγάλο βαθμό εκείνη η αγροτική πολιτική και πρέπει να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Η ξύπνια ανάπτυξη. Πρόκειται για μια σειρά επενδύσεων που γίνονται για την καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων, για την καλύτερη ενσωμάτωση των ερευνητικών πορισμάτων και για τη μεγαλύτερη καινοτομία. Εδώ υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Επίτροπο που ασχολείται με τα θέματα έρευνας για να μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερη ενσωμάτωση στον τομέα της γεωργίας και τον τομέα της αγροτικής μεταποίησης, των αποτελεσμάτων της έρευνας που μπορούν να βοηθήσουν καλύτερη ανταγωνιστικότητα και βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων. Για τους μικρούς γεωργούς, τι θα γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει να κατευθύνουμε τις άμεσες επιδοτήσεις όχι μόνο στην υποστήριξη του εισοδήματο, αλλά και ως μοχλό τροποποίηση των αγροτικών προοπτικών σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο στις περιοχές που υπάρχουν πληρωμές μέσω του δεύτερου πυλώνα για την προστασία του περιβάλλοντο, αλλά για το σύνολο του ευρωπαϊκού Εδάφου να τροποποιηθούν οι αγροτικές πολιτικέ για να υπάρχει και καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Αυτό είναι και ο στόχο μα. Οι άμεσε πυλωμέ να υποστηρίζουν μεν το εισόδημα των γεωργών, αλλά να βελτιώνουν και τι αγροτικέ πολιτικέ όλων. Και για τους μικρούς γεωργούς <clears throat> ο εξυγχρονισμός έχει αυτό το στόχο διευκολύνει την υποστήριξή τους και τους δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία. Και με τον τρόπο αυτό μπορούν να έχουν πιο άμεση πρόσβαση στις αγορές, πιο ε, εύκολη σύνδεση με τους καταναλωτές και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Αυτό δίνει λοιπόν στις μικρές επιχειρήσεις καλύτερη διέξοδο στην αγορά που μπορούν να βοηθηθούν από αυτή και αυτό περιλαμβάνει και τι οργανώσει ε, παραγωγών. Για το γαλακτοκομικό τομέα, παραδείγματο, χάρη, η πρότασή μα έχει σαν στόχο να ενισχύσει την διαπραγματευτική ικανότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων και παραγωγών. Αναφέρθηκε επίσης από τον κύριο Άσχοθ το θέμα της μεταρρύθμισης που το παρουσίασε, παρουσίασε τη μεταρρύθμιση σαν κενή πνεύματος καινοτομία για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Εγώ όμω θέλω να συζητήσω μαζί σα όλα αυτά τα θέματα για να σα δείξω ότι πράγματι έχει ένα όραμα η μεταρρύθμιση αυτή που αρθρώνεται γύρω από τρει στόχου. Να πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι τρεις στόχοι στους δύο πυλώνες της κοινή αγροτικής πολιτικής και επίσης και στις δύο ομάδες χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι παλιέ τις παλιές χώρες και τις νέες χώρες, όπου πρέπει να προσαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα όραμα μια Ευρωπαϊκή Γεωργία που δεν θα είναι μονάχα ανταγωνιστική, αλλά ανταποκρίνεται και στι προσδοκίε των πολιτών σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και του φυσικού πόρου και τη χωροταξική ισορροπία. Αυτά προς το παρόν λοιπόν και για το θέμα των μεταλλαγών που είναι απαραίτητοι για να είναι απαραίτητε για να είναι πιο αποτελεσματική η κοινή αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται καλύτερη χρήση του δημοσίου χρήματο για να συνδεθεί η οικονομική πτυχή με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, καλύτερη διανομή και κατανομή των αγροτικών πόρων μεταξύ κρατών μελών και περιοχών, μια μεγαλύτερη εστίαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την ανταγωνιστικότητα. Ο στόχος μας είναι να προσπαθούμε να επιτύχουμε έτη περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν την προσθέμενη αξία στον αγροτικό τομέα και νομίζω ότι έχω απαντήσει εν μέρη ή πλήρω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα που με απασχολεί και εμένα αλλά εν πάση περιπτώσει θα το θέσουμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Πρόκειται για τι ε, επιστροφέ εξαγωγών. Αυτό είναι ένα θέμα που με καίει και μέχρι τώρα δεν είπατε τίποτα επ' αυτού. Τώρα λοιπόν ε, θα διαβάσω τα ονόματα ε, των ομιλητών που έχουν στήσει το λόγο. Γένσεν Δαντά, Ια, Δόφμαν, Μπέαμαν, Σικιάσκι, Καπουλασάντος, Λάιν, Παουλσεν, Βόγε, Ρόντουστ, Βοητσιεχόφσκι, Γετζεγεύσκα. Αυτοί λοιπόν έχουν στήσει το λόγο. Ο Τζάνι. Πολύ σύντομα πολύ σύντομα να απαντήσω στην ερώτησή σας με έναν και μόνο αριθμό. Το 2010 χρησιμοποίησαμε 1% του προπολογισμού τη ΚΑΠ για τις ε, ε, επιστροφές των εξαγωγών. Μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αν θέλετε, όμως πριν από 10-15 χρόνια μιλούσαμε για ποσοστά άνω των 10% του συνολού του προπολογισμού για τι επιστροφέ των εξαγωγών. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει πέρσι να χρησιμοποιήσουμε μόλι, 1%. Έχουμε λοιπόν πλέον άλλα μέσα για να λύνουμε αυτά τα προβλήματα χωρί αρνητικό αντίκτυπο στη γεωργία των άλλων χωρών. Και ένα άλλο στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χώρα λεωμελητή που εισάγει τα περισσότερα προϊόντα των χωρών του Τρίτου Κόσμου, των χωρών του Νότου, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και η Ιαπωνία μαζί. Άρα, νομίζω η ευρωπαϊκή αγορά όχι μόνο έχει μειώσει τον αρνητικό τη αντίκτυπο στι τρίτε χώρε, αλλά είναι περισσότερο ανοιχτή από όλε τι υπόλοιπε ω αγορά για τα προϊόντα που έρχονται από τον Νότο. Ευχαριστώ. Εντάξει λέει η Πρόεδρος, ας το λάβουμε αυτό ως ένα θετικό μήνυμα ότι το 1% ε, δαπανάται για τις επιστροφές εξαγωγών αλλά ε, ας θεωρήσουμε ότι από το 2013 και μετά τίποτα, 0,0 θα είναι το ποσοστό που θα προβλέπεται για τις επιστροφές των εξαγών. Ο Τζάνι Λαβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι ορισμένα θέματα εξετάστηκαν ήδη ε, και στην ε, ανακοίνωση του Επιτρόπου για τη μεταρρύθμιση της κοινή Γεωργικής πολιτικής. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία έχουμε ήδη εξετάσει στο πλαίσιο της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Θα ήθελα βέβαια να αποδώσω ιδιαίτερη σημασία στην κοινή γεωργική πολιτική. Στις εργασίες αυτής της Επιτροπής εξετάσαμε τη διάρκεια του ε, πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και θα ήθελα λιγάκι να σκεφτούμε την διάρκεια αυτή σε, σχέση, σε άμεση σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί σε μία περίοδο όπου υπάρχει έλλειψη κονδυλίων, ε, θα πρέπει τα κονδύλια να τα χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας. Η εμπειρία που έχουμε κάνει μας έχει οδηγήσει στο να πιστέψουμε ότι ε, υπάρχει κάποια ασάφεια όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων και περάσουν ακόμα κάποια χρόνια μέχρι αυτά να εφαρμοστούν. Η ανάλυση των ε, δαπανών μας οδηγεί στο να σκεφτούμε πώς στις ε, περιόδους προγραμματισμού που προβλέπονται θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα κονδύλια έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική και βέλτιστη χρήση των κονδυλίων αυτών. Εάν λοιπόν κληθούμε να επιλέξουμε ίσως ένα συντομότερο χρονικό διάστημα για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο τότε θα υπάρχει κίνδυνος να προβάλλουμε τα αρνητικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος μέσα σε αυτό το πολιτικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου θα καταστεί δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο του ε, φιδελού αυτού πορού η ε, εισήγηση που παρουσιάστηκε εξαιρεί αυτά τα πέντε έτη του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να επιλέξουμε είτε τα επτά χρόνια είτε τα πέντε συν πέντε στην περίπτωση κατά την οποία ο προγραμματισμός επιτρέπει να έχουμε μια δεκαετή περίοδο προγραμμάτων και μετά να εξετάσουμε άλλα στοιχεία, όχι αυτά που προβλέπονται στον προγραμματισμό, αλλά αυτά που θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα διαχειριστεί κανείς σε ε, σε βάση. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στον, στη δομή του προϋπολογισμού. Ο εισηγητής μας μας παρουσίασε τρεις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Η μία λύση αφορά κυρίως ε, την διάρθρωση του προϋπολογισμού επί τη βάση της στρατηγικής 2020. Η άλλη εναλλακτική λύση αφορά τις ιστορικές πολιτικές και μια τρίτη εναλλακτική λύση ε, κατ' ουσίαν είναι εκείνη που λέει να διατηρηθεί η τρέχουσα δομή του προπολογισμού έστω και αν υπάρχει αυτή η έλλειψη πόρων, έστω και αν έκαναν αυτές οι αρνητικές εμπειρίες σε σχέση με την ευελιξία. Εγώ λοιπόν προφανώς θα πρέπει να διατηρήσουμε την τρέχουσα δομή του προϋπολογισμού και να υπάρχει μια κατάλληλη μια κατάλληλη γραμμή που θα προβλέπει την κοινή γεωργική πολιτική η οποία όμως αυτή θα είναι μόνη της, θα είναι απόλυτα διαχωρισμένη από τις υπόλοιπες. Ευχαριστώ η Μέρι Ριντ. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά από τα σημεία που ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη εγερθεί. Θέλω να είμαι σύντομη και θα μιλήσω μονάχα για ένα συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει κάποιο χαρακτήρας μυρολατρείας στην αντιμετώπιση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής και της μεταρρύθμισής της. Ε, ελπίζω να μην παρακολουθούν οι αγρότες από το διαδίκτυο τα λεγόμενά μας. Ελπίζω ότι είναι καλύτερο ο καιρό εκεί που βρίσκονται και είναι μαζί με τις αγελάδες και τα σπαρτά τους. Ένας από τους στόχους της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής που αφορούσε τα εισοδήματα των αγροτών δεν έχει πραγματοποιηθεί. Θα ήθελα να το αναγνωρίσει αυτό η Κομισιόν και να μας εξηγήσει πώς θα πετυχαίναμε κάποτε αυτούς τους στόχους που υποστηρίζουμε όλοι και που είναι γεγραμμένοι και στις συνθήκες. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Επίτροπο. Χαίρεται να διευθύνει μια πολιτική ένας από τους κύριους στόχους στους οποίες δεν έχει επιτευχθεί. Οι ίδιες οι στατιστικές της Κομισιόν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες σας που μας, τους, μας τις δίνουν, δείχνουν ότι οι άμεσες πληρωμές είναι ζωτικές για τους γεωργούς, ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος πολλών γεωργών. Γι' αυτό πρέπει να το θυμόμαστε αυτό όταν μιλάμε για την ενδεχόμενη μείωση της ε, υποστήριξης των γεωργών στον προϋπολογισμό. Αν δούμε τα πράγματα, αν σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα μυρολατρικά, πρέπει να σκεφτούμε και το ρόλο των αγορών. Έχουν αναφέρει πολύ την διαπραγματευτική ικανότητα των γεωργών στην αγορά των τροφιμικών προϊόντων. Η Κομισιόν δεν έχει δείξει να θέλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το πρόβλημα αυτό. Γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει και την πολιτική ανταγωνισμού που η δική μου εντύπωση είναι ότι εάν είναι φτηνότερα κάποια τρόφιμα δεν μας νοιάζει με ποιο τρόπο έχουν γίνει τόσο φτηνά. Θα πρέπει η Κομισιόν όμως να αντιμετωπίσει και την ηθική πτυχή της αγοράς τροφίμων. Έχουμε ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που μιλάνε για ηθική στον τομέα τον ε, τραπεζικό πιστοτικό, όπου σε μεγάλο βαθμό δεν υπήρχε αυτή η ηθική. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ίδιο πρόβλημα στον τομέα της γεωργίας. Έρχομαι τώρα στο επόμενο σημείο που αφορά το, την έννοια του δημόσιου αγαθού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να δούμε από μια άλλη οπτική γωνία, εγώ νομίζω, τα δημόσια αγαθά και ίσως μπορείτε να μου δώσετε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Μπορείτε να βρείτε ποιο είναι το αντίτιμο αυτών των δημοσίων αγαθών αν έπρεπε να γίνονται από δημόσιους υπαλλήλους. Πόσο θα κόστιζαν οι διακοπές για καφέ, οι προστατευτικοί εξοπλισμοί, οι διακοπές τους, όλα αυτά τα πράγματα, εάν έπρεπε δημόσιοι υπάλληλοι να ασκούν τη γεωργία και όχι γεωργοί που το κάνουν πολύ φτηνότερα. Αν λοιπόν όλα αυτά τα δημόσια αγαθά η προστασία του περιβάλλοντος, παραγωγή τροφίμων γινόταν από δημόσιους λειτουργούς και όχι οι αγρότες που το κάνουν σήμερα και δεν ζητούν το αντίτιμο αυτών των υπηρεσιών, τι θα μας κόστιζε τελικά μια τέτοια πολιτική. Νομίζω θα κόστιζε κάτι το αστρονομικό. Γι' αυτό, άμα το σκεφτεί αυτό κανείς, δεν θα πρέπει να ζητά περικοπή του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη επίσης και την ισοδίκια μεταχείριση υπάρχουν μεγάλες ανισο, ανισότητες μεταξύ των γεωργών. Είναι κάτι που το δεχτήκαμε όταν έγινε η συμφωνία για τη διεύνυση. Πρέπει όμως να υπάγεται, να υπόκειται και σε κάποια λογική αυτή η ισότητα. Μήπως θα πρέπει ο κάθε γεωργός να έχει την ίδια χρηματοδότηση. Όχι βέβαια, δεν είναι λογικό. Πρέπει να βρούμε μηχανισμούς να συνδέουμε αυτές τις πληρωμές με τους γεωργούς που είναι πραγματικοί ενεργοί γεωργοί και αυτό σημαίνει πιο σαφείς ορισμούς από ό,τι έχουμε σήμερα. Και κλείνω γιατί τελειώνει και ο χρόνος μου σε ό,τι αφορά τα θέματα εδαφικής συνοχής και προστασίας. Το υποστηρίζουν πολλοί από εμά. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε ένα σωστό εισόδημα στους γεωργούς, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα εδαφικής συνοχής ή της διατήρησης των φυσικών πόρων γιατί αλλιώς οι γεωργοί θα προσπαθήσουν να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους και να τις κάνουν πιο βιομηχανικές και θα χάσουμε γεωργού, θα χάσουμε την πυκνότητα πληθυσμού που είναι απαραίτητη σε μειονεκτικές περιοχές. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι χρήσιμο λοιπόν που έχουμε τη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να είναι λιγότερο φαταλιστική και μυρολατρική και πιο ρεαλιστική για όλους από εμά οι οποίοι μας ακούνε, εάν μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για αυτήν την Επιτροπή να είμαστε ρεαλιστέ στι προτάσει που θα κάνουμε και με τι διάφορε εκθέσει μα. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητάμε το θέμα αυτό σήμερα, διότι εγώ πιστεύω ότι ακολουθούμε ακριβώ αυτή την ρεαλιστική προσέγγιση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με του πόρους μας και πώς ακριβώς θέλουμε να θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Ε, για την ώρα, ε, στο έγγραφο που έχουμε, διερωτώμεθα αν θα παραμείνουμε στην ε, ίδια ιδέα που είχαμε το 2004 για συγχρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα. Χαίρομαι ιδιαίτερως για αυτό που είπε ο Επίτροπος. Βεβαίως, εάν υπάρξει συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνει αυτό ο τομής του προπολογισμού που έχουν βάρος, βαραίνει ο λόγος των κρατών μελών. Ε, για τα προγράμματα που θα συγχρηματοδοτηθούν. Αυτό δεν είναι περίπτωση του πρώτου πυλώνα που είναι ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πολιτισμού. Είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό κατά μέρο νομίζω. Όμως αυτό που θέλω να πω στον Επίτροπο είναι ακόμη μαζί μας είναι ότι συνεχίζω να πιστεύω ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η ιδέα σας στο να επικεντρωθούμε περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία είναι κάτι που θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Ναι, θέλουμε να εξυγχρονιστεί η γεωργία, να προχωρήσει, να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον. Διότι έτσι ε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής. Διότι θα μπορούμε να επικαλεστούμε την ε, πρόοδο. Ε, στον πρώτο πυλώνα κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τις πληρωμές που γίνονται για ιστορικούς λόγους. Θα πρέπει αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, θέλω να επεκταθώ λίγο σε αυτά που είπε ο κ. Σάσφορντ για την ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας. Είπατε ότι θέλατε δημιουργήσει συνάντηση με τον κύριο Άσφορντ για να το εξηγήσετε πώς λειτουργεί αυτό. Και εμείς θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τι θα λέγατε μεταξύ σα. Γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν συνεχίζει να κάνει μόνο όσα ξέραμε ω τώρα, αλλά πραγματικά δίνει ε, αποτελέσματα με μια πιο σύγχρονη αποτελεσματική γεωργία. Παρακαλώ. Κύριε Νταντά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ε, οι θεμελιωτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιούργησαν την αγροτική ε, πολιτική για την οποία μιλούμε σήμερα, θέλησαν να δημιουργήσουν και μια κοινή επιστημιστική πολιτική. Η πολιτική αυτή ήταν στατική σημασία, διότι ήταν καθοριστική για την ζωή, την επιβίωση των πολιτών μα. Δεν πρέπει να το αμελούμε αυτό. Επί 15 χρόνια μιλάμε συνεχώ για αγορά. Εγώ λοιπόν θέλω να επιγραμμίσω ότι στου νέου προσανατολισμού που μα παρουσίασε ο Επίτροπο, ε, βλέπουμε ένα νέο θεμελιώδη στόχο, ότι θα γυρίσει η κοινή αγροτική πολιτική στον πρώτο τη στόχο, τον ε, πρωταρχικό τη αυτό στόχο, να ταΐζει τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν προδιαγραφέ που δημιουργήθηκαν ε, με το πέρασμα των ετών στην Ευρώπη. Και έχουμε παραγωγή που ε, δίνει προϊόντα με την υψηλότερη ποιότητα παγκοσμίω λόγω ακριβώ των προτύπων που έχουμε θέσει. Εάν υπάρχει λοιπόν μια πρώτη αιτιολόγηση των βοηθειών που δίνουμε στου γεωργού, πρώτα απ' όλα είναι η ανταμοιβή για το επιπλέον κόστο που καλύπτουν λόγω των δικών μα των κανόνων. Α δούμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται σήμερα για να, προσ... να προσπαθήσει ο καθένα να κερδίσει προ τη θεμενή αξία και τι γίνεται με κάποιε τιμέ λόγω χάρη στην κτηνοτροφία. Βλέπουμε μια, έναν αγώνα δρόμου ε, για την παραγωγή που Κάποιες φορές όμως προκαλεί ατυχήματα όπως έγινε τώρα στη Γερμανία με τις διοξίνες. Όμως αυτή η πορεία, ε, αυτός ο αγώνας δρόμου θα μας οδηγήσει σε καταστροφές και θα παρεμποδίσει τους στόχους που θέλουμε να επιδιώξουμε. Πρέπει λοιπόν ω προ τον προλογισμό να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να καλύπτεται η γεωργία. Αυτό είναι σίγουρο όμω. Δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και του φραγμού που εμεί οι ίδιοι δημιουργούμε στην γεωργία. Διότι αν δεν λάβουμε υπόψη το σύνολο αυτό των επιπλέον υποχρεώσεων, συλλογικώ δημιουργούμε δυσκολίε στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, όχι μόνο στη γεωργία τη μια τη άλλη χώρα που ενδεχομένω παράγει περισσότερο από την άλλη. Να λοιπόν που ήθελα να σταθώ. Ε, αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, αλληλεγγύη μεταξύ των γεωργών και το ζήτημα της νομιμότητας της στήριξης. Νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι να οδεύσουμε προς την ισότητα της στήριξης. Όμως τι ισότητα θέλουμε, απόλυτη ισότητα μεταξύ των χωρών ή ισότητα ανάλογα με το μέσο εισόδημα των κατοίκων ή ισότητα ανάλογα με το μέγεθο του άκου που έχει αναλάβει κάθε χώρα. Διότι όταν θέλουμε να ενοποιήσουμε το εισόδημα, το μέσο εισόδημα των κατοίκων κάθε χώρα, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ε, ε, εξισορροπηθεί, να ε, είναι ίσο το βάρο που έχουν επομιστεί όλοι του. Ιδάλω δεν μπορούμε να έχουμε ισορροπή μεταχείριση όλων των χωρών μεταξύ του. Και επίση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία που έχει δημιουργηθεί, τίθεται και το θέμα των τιμών, τη ρύθμιση των τιμών και των αγορών. Ε, Αυτή την ιδέα την έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια, από την πλευρά τουλάχιστον τη Επιτροπή. Ο Επίτροπο το επεξεργάζεται, μα είπε. Έχει αναθέσει μελέτε για να εξευρεθούν νέε ιδέε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρί χρήμα, βεβαίω. Καταλαβαίνω και σημειώνω ότι τα κονδύλια γίνονται όλο και λιγότερα. Εάν λοιπόν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο εντό οποίο εργαζόμαστε, θα πρέπει να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, να τα βάλουμε κατά, κατά μέρο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα έτη των παχιών αγελάδων για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ισχνότερων ετών. Ε, και κάτι άλλο που μου φαίνεται σημαντικό. Αν θέλουμε να έχουμε μια ανιθάλια συζήτηση για τα θέματα των προπολογισμού και των πόρων τη Γεωργία, θα πρέπει επίση να σκεφτούμε τι γίνεται σε καθένα από τα κράτη μα. Να συγκρίνουμε το τι έχουμε λάβει σε σχέση με το τι δίνουμε. Γιατί εδώ χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να συζητήσουμε του ίδιου πόρου μεταξύ μας για να δούμε πόσο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον προπολογισμό μας. Ένας προπολογισμός που είναι προπολογισμός όλων, όχι προπολογισμός ενός εκ μέρους μας για τους υπολείπους. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Επίτροπο να μας ε, απαντήσει, διότι η ώρα είναι περίπου 11 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώ <clears throat> με το σχόλιο του κυρίου Λαβία για το μήκος της περίοδου προγραμματισμού. Είναι σαφές ότι ιδιαίτερα για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πέντε χρόνια είναι πολύ λίγα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται χρόνος εκπόνησης των προγραμμάτων, χρειάζεται διαπραγματεύσει με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα πολλές φορές σε κράτη-μέλη και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία πληρωμών. Νομίζω ότι πέντε χρόνια είναι πολύ σύντομος χρόνος και αυτό θα θίξει την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Υπάρχουν βέβαια πολλές επιλογές στη συνέχεια. Η Κομισιόν θα εκφράσει την απόψή της για την ε, ανακοίνωση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Νομίζω ότι ένας ε, χρονικός ορίζοντας 7 με 10 χρόνια από τη δική μου οπτική γωνία είναι μια καλύτερη χρονική περίοδος. Όσο πιο μακριά είναι αυτή η χρονική περίοδος, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Όπως είπε και ο Στεφάν Λεφόλ, χρειάζεται όταν πρόκειται για συμβατικά προγράμματα να υπάρχει αρκετός χρόνος. Σε ό,τι αφορά τη διάθεση του προϋπολογισμού, εγώ πιστεύω ότι επιχειρηματολόγησα και έδωσα στοιχεία λέγοντας ότι ήδη στους δύο πυλώνες της η κοινή αγροτική πολιτική έχει ένα συντονισμένο χαρακτήρα. Μια τεχνητή διαχω... Ένας τεχνητός διαχωρισμός των δύο πυλώνων στον προϋπολογισμό θα θίξει αυτή τη συνοχή και συνεκτικότητα που υπάρχει. Γιατί ο δεύτερος πυλώνας <clears throat> δεν αντιμετωπίζει μονάχα το θέμα της εδαφικής συνοχής. Αντιμετωπίζει και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Με ρωτήσατε πώς ο δεύτερος πυλώνας με όλες τις επενδύσεις εξυγχρονισμού, τις επενδύσεις κατάρτισης, δημιουργίας νέων προϊόντων, καινοτομίας. Όλα αυτά τα εργαλεία λοιπόν που αναφέρθηκαν το να υπάρχει κεφαλαιοποίηση στα καλά χρόνια για να καλυφθούν οι απώλειες στα δύσκολα χρόνια, όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ε, συμπληρωματικότητα μεταξύ των πυλώνων, να έχουμε μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση στους δύο πυλώνες και συγχρόνως μια ειδική αντιμετώπιση που λαμβάνει υπόψη να, λάβουμε, <clears throat> να αντιμετωπίσουμε την ε, ποικιλομορφία στα κρατημέλη και στην κατάσταση των γεωργών και στους δύο πυλώνες. Στην κυρία Μακίνες, έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και στο παρελθόν, συμφωνώ μαζί σας αν δούμε τα στοιχεία τα σημερινά, οι στόχοι της συνθήκης που έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ένα σωστό εισόδημα για τους γεωργούς δεν έχουν στην πράξη επιτευχθεί. Ακριβώς γιατί με όλες τις προδιαγραφές, με όλες τις απαιτήσει που υπάρχουν για τους γεωργούς έναντι των φορολογουμένων και των ε, καταναλωτών, υπάρχει μεγάλη πίεση για τους γεωργούς. Εξάλλου υπάρχει άνοιγμα των αγορών σε προϊόντα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν σέβονται πάντα τους κανόνες παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει θίξει το εισόδημα των γεωργών και κυρίως έχει διατηρήσει και οξύνει την ανισοκατανομή εισοδήματος μεταξύ των γεωργών. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι η απώλεια εισοδήματο των γεωργών λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής που έλκεται από τις αυστηρέ προδιαγραφές που θέτουμε στους γεωργού για την παραγωγή, αυτό το θέμα δεν μπορεί να λυθεί μόνο με την κοινή αγροτική πολιτική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι χρειάζεται μια διαφορετική κατανομή της προσθέμενης αξίας στην τροφιμική αλυσίδα η Κομισιόν δεν είναι αλήθεια ότι δεν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα όχι μόνο γεωργία, αλλά και βιομηχανική πολιτική εσωτερική αγορά ανταγωνιστικότητα. Και έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα φέτο στην Κομισιόν για μέτρα που πρέπει να ληφθούν από διάφορου επιτρόπου για το συγκεκριμένο αυτό ερώτημα. Ε, σίγουρο ότι μια καλύτερη κατανομή των ε, επιδοτήσεων και μια Ισοδίκια μεταχείριση δεν σημαίνει μαθηματική ισότητα των επιδοτήσεων, γιατί έχουμε διαφορετικές συνθήκες παραγωγής. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για την κατανομή των ε, επιδοτήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε ακόμα ιστορικές αναφορές κατά αγροτική εκμετάλλευση και κατά περιοχή στα παλιά κρατημέλη, αλλά δεν υπάρχει αυτό στα νέα κρατημέλη γιατί εισήλθαν μετά από τη μεταρρύθμιση του συστήματο αμέσων πληρωμών το 2003. Ο στόχο μα τώρα είναι να αντιμετωπίσουμε το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ίδια κριτήρια, αλλά η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων θα πρέπει να λάβει υπόψη και την διαφορά που υπάρχει μεταξύ αγροτικών εκμεταλλεύσεων και περιοχών, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια ισοδίκαια μεταχείριση αντιμετωπίζοντα καταστάσει διαφορετικέ. Για μένα αυτό σημαίνει μια δίκαια αντιμετώπιση. για τη συγχρηματοδότηση στον πρώτο πυλώνα. Δεν έχω να κάνω σχόλια. Συμφωνώ μαζί σας πλήρως. Το είπα ήδη προηγουμένως. Για το θέμα της ανταγωνιστικότητας νομίζω ότι απήντησα ήδη. Στον πρώτο πυλώνα αυτό αντιμετωπίζεται με τις άμεσες επιδοτήσεις. Και οι άμεσες επιδοτήσεις έχουν συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργών γιατί οι γεωργοί μας πρέπει να αντιμετωπίσουν γεωργούς από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τους αυστηρούς κανόνες των δικών μας γεωργούς. <clears throat> Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν τις ίδιες προδιαγραφές και τις ίδιες προϋποθέσεις, αλλά να κρατήσουμε και την ανταγωνιστικότητα των γεωργών. Ένα περαιτέρω στοιχείο είναι αυτό της επιδότησης για την ε, ποικιλομορφία των προϊόντων, για την ανταγωνιστικότητα και για την καλύτερη κατάρτιση των γεωργών μας. Θα πρέπει λοιπόν οι γεωργοί να ακολουθούν τα μηνύματα των αγορών, κάτι το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο τώρα με τη μείωση των τιμών εγγύησεως για τα αγροτικά προϊόντα. Αλλά παράλληλα πρέπει να έχουμε και τα εργαλεία τα οποία θα εξορροπήσουν καλύτερα τη ζήτηση με την προσφορά. Αλλά μπορώ να πω ότι για μένα είναι πιο ανταγωνιστική πια η ευρωπαϊκή αγορά θα εισάγουμε και νέα στοιχεία τα οποία θα θέλουν να διατηρήσουν το εισόδημα των γεωργών αλλά επίσης και τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Να υπάρχουν αμοιβαία ταμεία και εγγύηση εισοδήματος για τους γεωργούς ώστε να χρηματοδοτούνται από τους γεωργούς όταν είναι υψηλέ τιμές αλλά να αντισταθμίσουν την, την απώλεια εισοδήματος όταν πέφτουν οι τιμές και ανέφερα επίσης και την ενσωμάτωση των πορισμάτων της έρευνας στη Γεωργία. Αυτό θα είναι το οδηγό νήμα σε όλα τα μέτρα για καλύτερες επενδύσεις, εξυγχρονισμό και καλύτερη κατάρτιση. Με την Επίτροπο Έρευνα συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό, ώστε η βασική έρευνα να αντιμετωπίσει αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα των γεωργών και στη συνέχεια θα δώσει τα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν και στην πράξη τα πορίσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων κάτι το οποίο προφανώς θα συμβάλλει και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών μας. Αυτά λοιπόν. Μπορώ να κλείσω εδώ. Για αυτά που είπε ο κύριος Δαντέν δεν έχω να κάνω σχόλια. Νομίζω ότι κατά τα άλλα έχω απαντήσει πλήρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι έχουμε δείξει όλοι μια σημαντική αυτοπιθαρχία και έχουμε προχωρήσει καλά με το χρόνο που είχαμε θεσπίσει για αυτή τη συζήτηση. Αν τώρα πρέπει να φύγετε, σας αποχαιρετούμε ήδη. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει να μείνουν εδώ γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειές. Ο επόμενος... Ναι. Εμείς είμαστε Επιτροπή Σούρε. έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια έκθεση και να τη συζητήσουμε. Η έκθεση αυτή φυσικά αναφέρεται και σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Επίτροπος, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν το λόγο το πράττουν μόνο για τον εαυτό τους και για τον Επίτροπο. Το πράττουν και έναντι των άλλων συναδέλφων και εμείς πρέπει να θεσπίσουμε τις προτεραιότητές μας και να μπορούμε να συζητήσουμε και μεταξύ μας και όχι απλώς να πούμε στην Επιτροπή τι περιμένουμε να πράξει η Επιτροπή. Επομένως νομίζω ότι και για τον επόμενο γύρο είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις των ε, ε, ομιλητών. Ο επόμενος ομιλητής είναι κάποιος ο οποίος έχει φύγει, μετά ακολουθεί και ο Ντότμαν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στον σύντομο αυτό χρόνο που έχω θέλω να αντιμετωπίσω ορισμένα σημεία, δύο ζητήματα τα οποία ανέφερε ήδη ο κύριος Σλαβία. Πρώτα απ' όλα, ποια θα πρέπει να είναι η διάθεση του προϋπολογισμού Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει μέσα στην Επιτροπή μας και όχι αυτή καθεαυτή η αγροτική πολιτική. Είναι απαραίτητο να πω ότι υπάρχει μια δομή η οποία είναι ήδη καινοφανής. Δεν είναι παραδοσιακή και επομένω δεν είναι χρόνος ακόμα να την ε, τροποποιήσουμε. Επίσης μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια και εδώ μια επιλογή 5 συν 5 χρόνια δεν θα ήταν ανόητη. Ξέρουμε ότι ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μας δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει σε κάποιο βαθμό όμως να συμβαδίζει και με την ε, χρονική ε, διάρκεια της ε, θητείας του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, που είναι πέντε χρόνια. Είναι απαραίτητο, όπως είπε επίση ο κύριος Επίτροπος, να καλμάρουμε κάπως το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Έχει μόλις ε, περατωθεί η τέταρτη μεταρρυθμίση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Οι γεωργοί δεν καταλαβαίνουν <clears throat> ποια τι να κάνουν, γιατί συνέχεια μεταρρυθμίζεται η πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, πρέπει να πω ότι μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία η γραμματεία της Επιτροπής ε, Γεωργίας και όπως είπε η, η πρόεδρος της Επιτροπής μας Ελπίζουμε ότι μετά από το 2013 θα καταργηθεί πλήρως η διαδικασία των εξωτερικών επιδοτήσεων, των επιδοτήσεων εξαγωγής. Αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο με χαροποιούν να τα ακούω. Μετά από αυτά που ελέγχθηκαν με τον κύριο Επίτροπο είναι ένα δεύτερο θέμα, το θέμα της ισοδίκαιας κατανομής. Και εδώ βρίσκω ενδιαφέρον αυτό το οποίο παρουσιάζεται στο έγγραφο αυτό της Επιτροπής Γεωργίας, όταν μιλάμε για ισότητα μεταχείρισης υπάρχουν μερικά κράτη τα οποία είναι υποχρεωμένα να δίνουν 40% των ε, χρημάτων τους στον ε, πρώτο πυλώνα και άλλα 95% σε αυτό τον, ε, στο δεύτερο πυλώνα συγκεκριμένα. Συγγνώμη. Επομένως δεν πρέπει να δούμε μονάχα ένα τομέα και ένα πυλώνα χωριστά, θα πρέπει να δούμε και τους δύο τομείς για ορισμένες ε, χώρες. Είναι νευραλικός λοιπόν ο πρώτος πυλώνας και αυτό δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Και για να κλείσω τώρα τις παρατηρήσεις μου, η συνοχή μεταξύ πολιτικής συνοχής και πολιτικής γεωργίας, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και συμφωνώ με τον κύριο Επίτροπο, θα πρέπει το ένα χέρι να ξέρει, να ξέρει τι κάνει και το άλλο χέρο κάνει, το άλλο χέρι κάνει, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να είμαστε κουλοί. Πρέπει να έχουμε δύο χέρια και να συνεχίσουμε να έχουμε και την περιφερειακή πολιτική και την αγροτική πολιτική και να δώσουμε την ίδια αξία και στις δύο αυτές πολιτικές. Οι δύο πολιτικές αυτές εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους, μπορούν να έχουν κοινά στοιχεία, μπορεί να υπόκειται σε κοινή στρατηγική, αλλά πρέπει να μείνουν χωριστές πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτό νομίζω ότι ο Επίτροπος Τσόλος μαζί με την ε, Επίτροπο Αλληλείας και με τον Επίτροπο Περιφερειακών Θεμάτων και τον Επίτροπο Κοινωνικών Θεμάτων ήδη προσπαθεί να το κάνει. Το είπε αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβατοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να είναι στον δυνατόν πιο αποτελεσματική και αποδοτική η λειτουργία των πολιτικών αυτών. Αγροτική ανάπτυξη, αλληλεία, περιφερειακή πολιτική, κοινή αγροτική πολιτική. Ο Τάις Μπέρμαν έχει τώρα το λόγο. Συγγνώμη που θα σας καλάσω λίγο την ατμόσφαιρα, αλλά Εάν η επιστημιστική ασφάλεια είναι ο πρώτο λόγο που θα πρέπει η κοινή αγροτική πολιτική να είναι προτεραιότητα, αυτό βρίσκω ότι είναι ένα λαϊκιστικό επιχείρημα. Στι σύγχρονε γεωγραφικέ περιοχέ τη Ευρώπη, οι γεωργοί έχουν ένα λαμπρό μέλλον, γιατί παράγουν όχι μόνο για την Ευρώπη στι εύκολε αυτέ περιοχέ, αλλά και για μεγάλα μέρη του υπόλοιπου κόσμου, όπου η καλλιεργήσιμη γη συρρυκνώνεται και αυτό ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει. Η επισητιστική ασφάλεια λοιπόν είναι ένα ζήτημα στι αναπτυσσόμενε χώρε, όπου ένα δι ανθρώπων δεν είναι βέβαιο ότι αύριο το πρωί θα έχουν να φάνε. Αυτό έχει να κάνει με τι κακέ επενδύσει στην ε, περιοχή τη υπαίθρου στι χώρε του, με την φιλελεύθερη θεώρηση των αγορών, που όμω απέτυχαν κάποιε φορέ στου γεωργικού τομεί, στι αναπτυσσόμενε ακριβώ χώρε. Και επίση με το πόσο παραμελούνται οι γεωργοί σε αυτέ τι χώρε. Η επιστημιστική ασφάλεια για μα δεν είναι καθόλου ζήτημα. Οι γεωργοί έχουν λαμπρό μέλλον. Θα παράγουν. Πολλοί γεωργοί δεν έχουν καμία επιδότηση, καμία στηρίξη στην Ευρώπη και παράγουν. Παράγουν γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση και ολοένα αυξάνεται. Το επιχείρημα αυτό είναι τελείω εσφαλμένο. Το επόμενο επιχείρημα, η φυσική πόρη, να σα θυμίσω ότι το ίμιση τη απόλυτη τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη οφείλεται στην εντατική καλλιέργεια και γεωργία την τελευταία δεκαετία. Κάτι πρέπει να αλλάξει λοιπόν στην κοινή αγροτική πολιτική, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ω προ την προστασία των φυσικών πόρων. Χρειαζόμαστε του γεωργού περισσότερο από ποτέ για να παράγουν τρόφιμα και μη τρόφιμα. Ενέργεια. Για την αντικατάσταση των ε, παραγόγων. Του χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, αλλά θα βρίσκονται εκεί. Το επιχείρημα ότι η ΚΑΠ χρειάζεται για να κρατήσουμε τους γεωργούς στην Ευρώπη είναι τελείως απατηλό. Δεν είναι σωστό. Θα παραμείνουν, θα είναι εκεί και θα έχουν και πολύ καλό μέλλον. Ε, έπειτα, η εδαφική συνοχή. Η οικονομία των γεωργικών περιοχών στην Ευρώπη καθόλου δεν εξαρτάται πλέον από τη γεωργία. Ακόμα και στη Γαλλία. Η γεωργία είναι ένα αμεληταίο κομμάτι της οικονομίας της υπαίθρου, η οποία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τις υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε βεβαίω του Γιώργου, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα τοπία, το υπαίθρο μα όπω είναι. Όμω η κοινωνία νομίζω ότι είναι πρόθυμη να, πληρωμη, να πληρώσει γι' αυτό, για να μείνει το σκάνι όπω έχει, ε, ο βορρά των κάτω χωρών όπω είναι. Είμαστε πρόθυμοι να καταβάλουμε το τίμημα για να πληρώσουμε τι υπηρεσίε που μα προσφέρουν ε, οι περιοχέ αυτέ. Γιατί οι Γεωργοί δεν θα πάρουν τόσο πολλά την αγορά, είναι σαφέ για τι επιδοτήσει στο εισόδημα. Όπω είπε πολύ σωστά η Μαρίτ Μαγκίνε, ε, εδώ αυτέ ω τώρα έχουν φανεί απολύτω ανεπαρκεί. Αν δείτε τι επενδύσει που χρειάστηκε να κάνουν οι Γεωργοί, παραλόγω χαμηλό παρέμεινε το εισόδημά του. Και οι επιδοτήσει στο εισόδημα δεν του βοήθησαν καθόλου όπω θα έπρεπε. Τουλάχιστον αυτό μα λέει το επιχείρημα αρχικά. Το μισό των ε, επιδοτήσεων αυτών ξεφεύγουν προ όσου πολλούν αγαθά προ του γεωργού και του ιδιοκτήτε των εδαφών. Τέταρτο σημείο, κοινή αγροτική πολιτική είχε καταστροφικές συνέπειες για τους γεωργούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό ε, σταματάει, πάβει και είναι ένα καλό στοιχείο αυτό. όπω είπε πολύ σωστά ο Επίτροπος, εισάγουμε περισσότερα ε, γεωργικά προϊόντα από τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες, περισσότερα από κάθε άλλη ήπειρο η παγκόσμια δύναμη. Και ε, σιγά σιγά επιδοτήσεις μειώνονται, απλώς δεν έχουν εξελιχθεί πλήρως. Όταν είχαμε τη γαλακτοκαιμική κρίση πριν από δύο χρόνια, αμέσω η Επίτροπο Φίσερμπελ χρησιμοποίησε το μέσο τη επιστροφή των εξαγωγών για να στηρίξει του ε, παραγωγού γαλακτοκομικών. Είναι κακή πολιτική αυτή και μπορεί να πάυσει. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να συζητήσουμε περισσότερο για την αναγκαία μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τη γεωργία, θα έχουμε γεωργού. Εγώ έχω απόλυτη πίστη σε αυτό. Εγώ του θαυμάζω, του εμπιστεύομαι. Χαίρομαι πολύ για τη δουλειά του, αλλά χρειαζόμαστε διαφορετική αγροτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα. Αν αυτά που λέμε για την κοινή αγροτική πολιτική την κάνουν να είναι πραγματικά μια κοινή αγροτική πολιτική, μια κοινή αγροτοπεριβαλλοντική πολιτική. Υπάρχει χώρος σε αυτή την πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχουμε προσθέσει νέα καθήκοντα στην κοινή αγροτική πολιτική. Ποιο είναι το αντίτιμο όμως αυτών των νέων καθηκόντων. Μήπως χρειαζόμαστε ένα νέο ορισμό του τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Να την ονομάσουμε κοινή αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική. Αν μιλάμε λοιπόν για μια νέα πολιτική και έχουμε στο μυαλό μας μονάχα τις παλαιές κατηγορίες και τους παλιούς ορισμούς, δεν λειτουργεί αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε και την οτροπία μας. Ο κύριος Επίτροπος είπε ότι το εισόδημα των γεωργών είναι το χαμηλότερο σε όλη την αγορά εργασίας. Μα τότε, παρά την γενεοδορία της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι τόσο χαμηλό το εισόδημα των γεωργών. Τελική ανάλυση. Πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά λοιπόν επιδοτείται ο καταναλωτής, επιδοτούμαστε όμως εμείς. Δεν φτάνουν τους παραγωγούς οι οποίοι πολλούν στους καταναλωτές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή μεταφοράς κονδυλίων και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη συνολική μας αξιολόγηση. Τέλος έχουμε και το πρόβλημα των αγορών γεωργικών τροφίμων. Ξέρουμε τι έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Υπάρχουν τεράστια κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κανείς δεν συζήτησε καν για αυτό το θέμα. Δημιουργήθηκαν οι απαραίτητοι φορείς για την εποπτεία των χρηματαγορών Υπήρξε μια σαφής παρέμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Όταν όμως έρθουμε στην Γεωργία, φαίνεται ότι ακολουθούμε τον Αδάμ Σμιθ για το αόρατο χέρι που διευθύνει και εξομαλύνει τις αγορές. Μα υπόκειται σε τόσο πολλές αβεβαιότητες η γεωργία, αν η συγκομιδή θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το προβλεπόμενο. Εάν δεν έχουμε πρόβλεψη και εξομάλυνση, οι αγορές θα καταρρεύσουν. Χρειαζόμαστε μία σωστή και πρόσφορη παρέμβαση στις αγορές. Όλοι φαίνεται να θέλουμε αυτή την παρέμβαση των αγορών, αλλά είμαστε ιδιαίτερα άτολμοι για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Τέλος. Θέλω να θέσω και το εξής ερώτημα. Έχουμε ανοίξει την αγορά μας στα προϊόντα τρίτων χωρών, ίσως υπερβολικά. Φαίνεται ότι εμείς δεν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε, να υποστηρίξουμε τις ε, χώρες αυτές. Αυτή τη στιγμή όμως ακολουθούμε λανθασμένη οδό και χρησιμοποιούμε λανθασμένα εργαλεία. Το τελευταίο ερώτημά μου είναι, θα έχουμε αρκετούς πόρους για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτά μας είπε ο κύριος Επίτροπος. Δεν αποτελούν υποστήριξη των περιοχών της υπαίθρου. Είναι ουσιαστικά θέματα πρώτου πυλώνα. Η πρασινοποίηση της οικονομίας, το πρασίνισμα της οικονομίας και οι επενδύσεις που επιδοτούνται Όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ καλά. Αλλά εγώ τολμώ να είπω ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν θα έχει τους απαραίτητου πόρους για να υποστηρίξει τη διαδικασία ανάπτυξης της υπαίθρου. Εμείς αυτό όμω θα πρέπει να υποστηρίξουμε και όχι τα αγροκτήματα αυτά κάθε αυτά. Μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστό αυτό που θα σας πω, αλλά το 2007 ξεχάσαμε πάρα πολύ σύντομα το ότι υπήρξε μια κρίση τροφίμων. Γιατί αυτή η κρίση παρέκαμψε την ε, Ευρώπη. Αλλά βλέπετε τον τρόμο στα πρόσωπα των, γεωργο... των ε, ε, πολιτικών όταν αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν σε περιπτώσεις κρίσης τροφίμων για να καλύψουν τις ανάγκες τη κοινωνία μα. Χρειαζόμαστε περισσότερη συζήτηση γιατί μιλάμε και για τη γεωργία και για το περιβάλλον και για τα τρόφιμα και τα τρόφιμα έχουν να κάνουν και με την υγεία και την ευμάρεια των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι από μόνοι του οι γεωργοί θα έχουν λαμπρό μέλλον. κάπω, πρέπει να τροποποιηθούν τα θέματα αυτά της παραγωγής τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρος. Ο Λουίς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ούτε. Ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους που δεν είναι μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρους, ιδίως τον συνάδελφο Μπέρμαν, ο οποίος μόλις έφυγε δυστυχώς, διότι τα επιχειρήματα που εκείνος χρησιμοποίησε είναι, θα μπορούσαν να είναι εύστοχα. Όμως εδώ μιλάμε για την κοινή αγροτική πολιτική που έχουμε όχι για αυτήν που θέλουμε όμως για το μέλλον. Καταλαβαίνω ότι εκείνος ε, αξιολογεί τα πράγματα έτσι επειδή είναι από την Ολλανδία ο κύριος Μπέρμαν. Όμως η Ολλανδία είναι προφανώς μια χώρα της Ευρώπης όπου ε, μπορεί κανείς να καλλιεργεί εδάφη χωρίς να υπάρχει καμία ρήπανση στα ύδατα. Όπου μπορεί να χρησιμοποιεί το ελάχιστο τετραγωνικό μέτρο γης που υπάρχει χωρίς καμία ρήπανση. Όμως η Ευρώπη δεν είναι σαν την Ολλανδία. Εάν θέλουμε μια γεωργία για το μέλλον της Ευρώπης, θέλουμε μια γεωργία όχι όπως έχει καλή αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στις κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν ε, η Γεωργία φαίνεται ότι σήμερα δεν ήταν ποτέ αναγκαία όσο μάλλον η γεωργία ποτέ δεν υπήρξε τόσο αναγκαία όσο σήμερα. η γεωργοί χρειάζονται στήριξη και η αστάθεια των αγορών ποτέ δεν υπήρξε τόσο σοβαρή. Ούτε έθεσε σε κίνδυνο την προμήθεια τροφίμων και των αγαθών ε, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λοιπόν τα τελευταία χρόνια απέχουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη ως προς την άνοιγμα των ε, Αγορώνουμε στα τα γεωργικά προϊόντα, διότι θέτουμε τεράστιες απαιτήσεις στους γεωργούς μας και από περιβαλλοντικής άποψης και από τις άποψεις της ευημερίας των ζώων. Έχουμε τις πιο απαιτητικές μεταρρυθμίσεις παγκοσμίω ως προς τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας προδιαγραφές. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα μέτρα στήριξης της αγοράς, διότι καταργούμε την στήριξη και τα άμεσα κίνητρα προς την παραγωγή. Από την άλλη διευρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλα δύο κράτη-μέλη και σχεδόν διπλασιάζουμε τον αριθμό των ε, γεωργών ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε δραστικά τον προπολογισμό μας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο χωρίς στηρίξει μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας δεν έχει καμία δυνατότητα να είναι οικονομικά βιώσιμη στο μέλλον. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καινούργια ΚΑΠ. Μια ΚΑΠ με νέο κύρος ε, και νέα νομιμότητα στο μέλλον. Θα πρέπει να είναι ένα μέσο υπεράσπισης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι ένα μέσο, μέσο ε, προστασίας της βιοπικιλότητας, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει η κοινή αγροτική πολιτική να είναι πηγή απασχόληση και υπεράσπιση τη εδαφική συνοχή. Οι γεωργοί στο μέλλον δεν θα πρέπει στο μέλλον να, να ασχολούνται μόνο με το τι ποσότητε θα παράγουν, αλλά να ε, καλύπτουν στο μέλλον να προσφέρουν μάλλον αγαθά προς την κοινωνία, ε, αγαθά τέτοια που τα χρειάζονται οι υπόλοιποι πολίτες. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να κρίνονται. Και η βάση των βοηθειών της ΚΑΠ θα πρέπει ακριβώς να λαμβάνει υπόψη και το κριτήριο της απασχόλησης στο μέλλον. Διότι το κριτήριο της απασχόλησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να κινητοποιήσουμε την παραγωγή και να νομιμοποιήσουμε μια πολιτική σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης οξίας, ε, που υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργία σε όλη την Ευρώπη, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου αυτό λοιπόν το λόγο ο προπολογισμό τη ΚΑΠ είναι απολύτω ε, θεμελιώδη σημασία. Θέλω εδώ να επισημάνω στου συναδέλφου ότι θα πρέπει ε, να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε την έκδοση Λάιον και τοποθετήθηκε προ το θέμα αυτό δεν θυμάμαι αν κατά 80-90% εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο η έκθεση αυτή. Αν θέλουμε λοιπόν ο προπολογισμό τη ΚΑΠ να παραμένει σταθερό δεδομένων των δυσχερών συνθήκων, θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και για το 2013 ήδη. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσω του συναδέλφου να είμαστε συνεπεί ε, και σε σχέση με το τι είπαμε στο παρελθόν και με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτή και για το μέσα του προπολογισμού που θέλουμε να αποδώσουμε για του στόχου μα. Είναι αναγκαίο αυτό. Θα πρέπει ο προπολογισμό να παραμένει στα επίπεδα αυτών που είχαν προβλεφθεί αρχικά Πρόεδρο, πολύ ωραία. Τώρα έρχεται επιτέλους ο εισηγητής, ο κύριος Λάιν. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ε, γιατί τα περισσότερα θέματα που ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη αναφερθεί. Καταρχήν να πω το εξή. Πάμε στη σελίδα 5 του εγγράφου της Επιτροπής ε, ΣΟΥΡΕ και αν δει εκεί κανείς ε, το γράφημα, το γράφημα δείχνει ότι εξετάζεται το όγκος του προϋπολογισμού της ε, ΚΑΠ και το ποσοστό που καταλαμβάνει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0,3 περίπου της 100. Η ΚΑΠ, όλοι είπαν, είναι η πιο κοινοτικοποιημένη πολιτική που έχουμε και αν το έχει αυτό κανείς ε, κατά νου καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό είναι ελάχιστο ε, και δεν έχει σχέση με αυτό ε, που δίδεται για την υγεία και την παιδεία που είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά. Αν δει κανείς άλλα γραφήματα, ας πούμε για την ΚΑΠ, το ποσοστό μειώνεται τα τελευταία 20 χρόνια από 80% έχει φτάσει στο 39,3%. Θα φτάσει το 39,3% το 2013. Βλέπουμε λοιπόν το πλαίσιο και την αναλογικότητα ε, υπάρχει εντωμεταξύ και η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά δεν προβλέπονται επιπρόσθετα κονδύλια για να ε, υλοποιηθούν κάποιες από τις προσδοκίες με αυτή τη νέα ε, συνθήκη που έχει τεθεί σε ισχύ. Δύσκολη λοιπόν η κατάσταση δημοσιονομική και αν ε, λάβουμε υπόψη μας και την επιστολή που εστάλει από τους πρωθυπουργού. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση. Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η ΚΑΠ δεν θα διονγκωθεί. Ε, μάλιστα ε, βλέπουμε ε, με την πάροδο των ετών ότι υπάρχει κάποια μείωση των κονδυλίων για την ΚΑΠ. Ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκομμένη ως ε, προς την στήριξη προς τους γεωργούς. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι ιδιαίτερα επιθετικοί ε, και ένας βασικός στόχος τους είναι να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν τις δικές μας τις αγορές. Εάν υπάρξουν υπάρξει σημαντική μείωση της υποστήριξης, καταλαβαίνετε ότι θα δώσουμε πεδίο δράσης ε, στους αντιπάλους μας. Και θεωρώ ότι ε, όλες οι αναπτυγμένες χώρες ε, πρέπει να πολεμήσουν για αυτό το θέμα στον ΠΟ. αλλιώς όπως σας είπα θα παραδώσουμε μερίδια της αγοράς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορούν στον προεπλογισμό και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημοσιονομικό θέμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των νέων κρατών μελών για μια πιο ισομερή κατανομή του προϋπολογισμού. Από το 2013 και μετά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ε, θα έχουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία από το 2013 και μετά. Ε, υπάρχει λοιπόν η ανάγκη καλύτερων, καλύτερης στοχοποίησης ε, θέσης πιο αποτελεσματικών στόχων. Η στατική 2020 είναι μια προτεραιότητα. Η αηφορία, η κλιματική αλλαγή, για μένα αυτά είναι θέματα κλειδί. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι παλιές ε, μέθοδοι καλλιέργειας που βασίζονταν στην ε, φτηνή ενέργεια, στο φτηνό πετρέλαιο, αυτές οι πολιτικές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για να καλύψουμε την ε, τεράστια αλματώδη αύξηση της ε, ζήτησης ε, που θα υπάρξει ε, από το 2013 και μετά η ασφάλεια των τροφίμων δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά όλο τον κόσμο και εδώ πρέπει να παίξει η Ευρώπη το δικό της ρόλο. Πρέπει εμείς να καλύψουμε τις ανάγκες ε, των ε, καταναλωτών μας. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι δυνατόν να καλυφθεί. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, να συμβαδίζει αυτή με την στρατηγική του 2020 και αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να παρουσιάσουμε, να μεταρρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων, ε, πιο αποτελεσματική χρήση. Και πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική και κοινέ αγορέ, Διότι μία από τι εύκολε λύσει ίσω να είναι η συγχρηματοδότηση. Αυτό μπορεί κανεί να το προτείνει ως ε, εύκολη λύση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση τη γεωρική πολιτική και τα κράτη-μέλη θα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για τι επιδοτήσει. Κάποια θα θέλουν, αλλά δεν θα θέλουν επιδοτήσεις. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία να διατηρήσουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή προσέγγιση. Αυτό σημαίνει καλύτερους στόχους και καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των υπαρχόντων πόρων. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο για να βάλετε τα ακουστικά σας και θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος ε, ε, Λάιν. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί μέσα στο πλαίσιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε χρήματα, υπάρχουν στενότητες προϋπολογισμού σε όλα τα κράτη-μέλη σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες που έχουν καλή χρηματοοικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση από τις άλλες, αλλά ο, η ευθύνη μας είναι να χρησιμοποιήσουμε με το πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο δυνατό τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας. Προφανώς θα χρειαζόμασταν περισσότερα χρήματα. προφανώς θα ήταν χρήσιμο να είχαμε μεγαλύτερο προπολογισμό. Αλλά αυτό είναι μια απλοποίηση των πραγμάτων θέτομεν το κεφάλι μας εντός της άμμου, όπως μία στουρθοκάμιλος, εάν έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε, όσο περιορισμένα και να είναι, για να μπορέσουμε να είμαστε στο ρετό πιο αποτελεσματικοί, ιδίω μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης των ζωνών της υπαίθρου. Πρέπει προφανώς να παραγάγουμε τρόφιμα, αλλά πρέπει παράλληλα όλο και περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε τη γη, τα δάση για να επιλύσουμε και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής. Οφείλουμε στα παιδιά μας να τους δώσουμε μια γη η οποία να στέκεται στα πόδια τους, να διατηρήσουμε το κλίμα, να διατηρήσουμε την βιοποικιλότητα. Θα πρέπει να κινηθούμε όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Ας είμαστε λοιπόν ριζοσπάστες. Γιατί ο πρώτος πυλώνας πρέπει να αφορά μονάχα την βοήθεια προς το εισόδημα των γεωργών. Γιατί δεν πρέπει να <clears throat> σκεφτούμε ορισμένα κράτη-μέλη, αυτά που έχουν καλύτερη ε, οικονομική κατάσταση, να δίνουν μεγαλύτερη συνεισφορά, 120% ενώ τα πιο φτωχά 80%. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισορροπία και θα δείχνει και μία αλληλεγγύη. Εντάξει, δεν πρέπει να ονειροπολούμε, αλλά είναι απαραίτητο να σκεφτούμε καλύτερα στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αλληλεγγύη των κρατών μελών. Και για το δεύτερο πυλώνα. Εδώ σας υπενθυμίσω ότι ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη για τα 70% των περιπτώσεων αφορά μονάχα 5 εκτάρια. Αυτές λοιπόν οι μικρές επιδοτήσεις μπορούν να έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, μπορούν να πάρουν τη βοήθεια για να επιδοτήσουν. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι οι κοινοί πόροι <clears throat> και τα κοινά μέσα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και την συσσωρευμένη από χρόνια εμπειρία στον αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να δούμε κυρίως πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των μικρών γεωργών οι οποίοι μπορούν να στραφούν σε προϊόντα ιδιαίτερα και να έχουν ανταγωνιστικότητα και εξαγωγική δυνατότητα σε <clears throat> προϊόντα ειδικών αγορών. Καταπληκτικά τυριά. Να βρουν μια ειδική θέση στην αγορά να παράγουν τα προϊόντα αυτά και έτσι θα έχουμε στην αγορά ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη της ιδιαιτερότητας παραγωγής και διανομής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 24 ώρες και μόνο έχει ημέρα. Δεν μπορούν οι γεωργοί να δουλεύουν περισσότερο και να παραγάγουν περισσότερο. Σιγά σιγά λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Και εδώ θέλω να σας τα πω. Γίνονται σήμερα επενδύσεις και υπάρχουν και άλλες επενδύσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για να εγκαθιδρύσουμε ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται σε δανειοδότηση με παροχή εγγύησεων όπως γινόταν τον παλιό καλοκαίρο. Αυτό θα μπορέσει να μας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία γιατί με τα δάνεια αυτά θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ατομική ευθύνη και μεγαλύτερη ελευθερία επενδύσεων από τους μεμενωμένους γεωργούς. Έτσι θα επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους μας. Όλοι πρέπει να τα σκεφτούμε λοιπόν αυτά τα θέματα και αυτές τις επιλογές Πρέπει να τολμήσουμε να είμαστε διαφορετικοί εν ώψη της τωρινής οικονομικής κρίσης που μας δίνει όλο και λιγότερες δυνατότητες. Μερσή, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ το βρήκα πολύ σωστό το ότι ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής που περιλαμβάνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί κατά την άποψή μου πολύ συχνά αγνοεί κανείς αυτούς τους στόχους της συζήτηση που γίνονται. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε και το είπε ο κύριος Λάιν ότι σε αυτή τη συζήτηση Οι μέχρι τούδε μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 20 ετών πρέπει να προβληθούν και να επενεθούν γιατί αυτές έφεραν δυναμισμό στη Γεωργία και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι διαδικασίες προσαρμογής που ακολούθησαν ήταν επιτυχείς. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στην ανακοίνωση της Κομισιόν εκείνο που δεν βλέπω να υπάρχει είναι το εξής. Ό,τι και να λέμε για το πρασίνισμα και για νέα στοιχεία που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και με τη συνεισφορά της γεωργίας, εκείνο το οποίο έχει σχέση με την cross compliance και εκείνο το οποίο ελέγχεται σήμερα και είναι απόλυτη προϋπόθεση για τις άμεσες πληρωμές, μα αυτό δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση Κομισιόν, τουλάχιστον όχι επαρκώς. Ε, αναφέρεται εν παρόντο Παρεπιπτόντος και όποιος δει το τι σημαίνουν αυτοί οι 20 κανονισμοί από την προστασία των, ε, του εδάφους μέχρι τον έλεγχο των λοιπασμάτων θα καταλάβει ότι ε, θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο επιθετικοί απέναντι στην Κομισιόν για να μην νομίζουν πολλοί ότι ξεκινάμε από το μηδέν. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι βεβαίως και στην όλη συζήτηση για τον προεπολογισμό για τη Γεωργία, το είπε αυτό και ο Επίτροπος, βεβαίως ε, θα πρέπει να γίνει συζήτηση το τι θα γίνει στις αγορές, τι θα γίνει για τους γεωργούς και τους καταναλωτές αν, αν δεν είχαμε αυτή την πολιτική τροφίμων που έχει άμεση σχέση με έμεση φορολογία. Πώ θα αντιδρούσαν οι αγορέ. ποιε θα ήταν οι επιπτώσει για του γεωργού ευρύτερα. Ίσως η Κομισιόν πρέπει να μα δώσει κάποια συγκεκριμένη στοιχεία. Ξέρω ότι υπάρχει το Ινστιτούτο Βάγκενινγκ, το οποίο μαζί με άλλα υπολόγισε ε, ή έκανε κάποιε προεκτάσει, κάποιε προβολέ ε, του τι θα σήμαινε Ποιε ήταν επιπτώσεις στα εισοδήματα όπως σας είπα αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική τροφίμων χρηματοδοτούμενη από τους φόρους και μια πολιτική η οποία στο παρελθόν οδήγησε σε σταθερότητα των τιμών. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι δεν υπάρχει αντίφαση μόνο με αυτά που ο κ. Μπέρμαν, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Το είπα και στην άλλη ο κ. Σικέρσκι. Κάναμε κάποιε εμπειρίε το 2007 με την κρίση των τροφίμων και τότε εκείνο το οποίο συζητήσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με άλλου διεθνεί οργανισμού οδήγησε στο ότι ο τότε επίτροπο είπε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την μέχρι μέχρι τώρα πολιτική ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν κάποια λάθη. Και πρέπει να συζητήσουμε και τι ε, επιδοτήσει ε, από τον προπολογισμό. Τότε εγώ ήμουνα ε, συνδιαπραγματευτή για το εργαλείο περί τροφίμων και διαπιστώσαμε ότι από τις πάνω από 75 χώρες οι οποίες από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο πήραν αναπτυξιακή βοήθεια λόγω της δομής ούτε καν 30 από αυτές δεν μπόρεσαν να διοχετεύσουν τα κονδύλια για την ασφάλεια των τροφίμων. Και μετά τι κάνουμε, ε, εκπλησόμεθα που αυτές οι χώρες δεν γίνονται αυτάρκες. Μα πρέπει καταρχήν να ξεκινήσουμε στην αναπτυξιακή πολιτική και να θίξουμε το θέμα των σωστών προτεραιοτήτων για τους πολίτες. Δεν νομίζω ότι γίνεται ικανοποιητικά κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή με και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περισσότερα τρόφιμα και πρώτε ύλε από αναπτυσσόμενες χώρες, από του Αμερικανούς, Καναδούς. Ε, τους Αυστραλούς ε, και τους Ιάπωνες, από ότι όλοι αυτοί μαζί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία πολύ προσεκτικά. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για δασμούς ή για μη δασμολογικά εμπόδια ε, τα οποία προβάλλονται πολλές φορές ε, ως τα πιο καθοριστικά. Και μετά υπάρχει και κάποια ιδεολογική προσέγγιση ανάμεσα στην ε, βιομηχανική γεωργία και τη γεωργία των μικρομεσαίων. Το να το κάνουμε αυτό, αυτό δεν νομίζω και δεν είναι σωστό, γιατί μας ε, αποσπά από ουσιαστικά προβλήματα. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα της ε, προστασίας του κλίματος, σε αυτόν τον τομέα χρειαζόμαστε έρευνα και τεχνολογική πρόοδο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίω, εγώ το λέω αυτό τώρα από τη δική μου την πρακτική εμπειρία, γιατί και εγώ ίδιο για 20 ολόκληρα χρόνια άρμεγα τη Αγελάδης και ε, η Αγελάδα των 20 ε, λίτρων είναι πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον από αυτή των 5 λίτρων. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η τεχνική αυτή δημιουργία αντιθέσεων δεν βοηθάει. Εκείνο που βοηθάει είναι το να θέσουμε στόχους. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την αηφορία, πώς μπορούμε τα δημόσια αγαθά για τα οποία ο Γιώργος δεν παίρνει καμία ικανοποιητική τιμή στην αγορά, να μπορούμε αυτά να τα στηρίξουμε και σε τελική ανάλυση πώς είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να θέσουμε αποτελεσματικότερους στόχους στην κοινή γεωργική πολιτική. Μέχρι σήμερα δεν δόθηκαν οι ικανοποιητικές απεντήσεις. Οι διακυμάνσεις των αγορών ε, τα επόμενα χρόνια θα μας δημιουργήσουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα. Ίσως ε, όχι τόσο ε, πρόβλημα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περισσότερο για χώρες όπου περίπου το 80% των εισοδημάτων πολιτών εξαρτάται από την ανέργεια. Αυτό που ενδιαφέρει επίση είναι και αυτό που διαφαίνεται τώρα ως τάση και σίγουρα έχει άμεση σχέση με την κερδοσκοπία. Κερδοσκοπία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καθήκον είναι διεθνέ για να υπάρξει μια κάποια σταθερότητα η οποία είναι απαραίτητη έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια αξιόπιστη και σταθερή, έναν αξιόπιστο και σταθερό εφοδιασμό με τρόφιμα. Γι' αυτό λοιπόν η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι κάτι το παροχημένο, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη και γενικότερα. Πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Και κλείνω ε, να πω κάτι σχετικά με τη διάρκεια της δημοσιονομικής πρόβλεψης, ε, της ευελιξίας και πώς είναι δυνατόν να ε, διαρθρώσει κανείς ένα προπλογισμό. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ε, προτείνω σε όλους να μην δεσμευτούν να μην έχουν προκαταλήψεις. Να πω το εξή. Όσο χειρότερα είναι τα στοιχεία, τόσο μικρότερη πρέπει να είναι η χρονική διάρκεια. Και αν είναι σωστά τα στοιχεία, εντάξει, α ισχύσουν και για 10 χρόνια. Και στην περίπτωση αυτή, η πρόταση προ το Συμβούλιο θα είναι, ξέρετε, διαπραγματευτείτε με το Κοινοβούλιο μόνο μία φορά τα 10 χρόνια και όχι δύο. Ίσως βοηθήσει αυτή η προοπτική. Αυτά λοιπόν όλα σχετίζονται. Κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Γεωργίας είναι υπέρ της μεγαλύτερης διάρκειας όπως και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στις επόμενες συνεδριάσεις. Κατανοώ βέβαια ότι χρειαζόμαστε σταθερό σχεδιασμό και όχι κάθε πέντε χρόνια να επιβάλλουμε στην Ευρώπη ένα νέο πρόγραμμα ε, κάποια προσαρμοστικότητα, συνέχεια και όχι κάθε πέντε χρόνια ε, καινούργια προγράμματα. Αυτό κανεί δεν μπορεί να το αντέξει. Αλλά ε, χρειαζόμαστε σε άλλου τομεί ε, και ευελιξία και κινητικότητα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι αυτά κάπω να τα συνδυάσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε. Και χρειαζόμαστε και αυτό ε, που υπόθηκε ότι αν υπάρχουν κάποια υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις ε, στους προπολογισμού. αυτό εντωμεταξύ το υποσχέθηκε ο Επίτροπο κ. Λεβαντόσκη να εξετάσουμε κατά πόσον αυτά τα τα υπόλοιπα θα μπορούμε από τη μία χρονιά να τα μεταφέρουμε στην επόμενη έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την ε, τεχνική αλλά απαραίτητη συζήτηση που έπρεπε να γίνει για τη διαμόρφωση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο. Το τελευταίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε όλοι μας. Αυτό ισχύει για όλες τις ε, πολιτικές και όχι μονάχα τις αγροτικέ πολιτικές. Η Ούλρικε, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω που σήμερα δώσαμε τόσο χρόνο για να συζητήσουμε δελεχώς το θέμα αυτό. Βλέπει από πολλέ παρεμβάσει κανείς ότι υπάρχει μια σχετική συνένεση για τον τομέα της γεωργικής πολιτικής και που υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές. Εγώ θέλω να εστιάσω περισσότερο στην ασφάλεια των τροφίμων και την διατήρηση τροφοδοσίας με τρόφιμα τα οποία είναι ποιοτικά υψηλή στάθμης αλλά είναι και προσβάσιμα και δυνατό να τα αγοράσει ο καταναλωτής. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ώστε το σύστημα των αμέσων πληρωμών να διαμορφωθεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε όχι μονάχα να έχει τη συνένεση των γεωργών αλλά συγχρόνως το σύνολο της κοινωνίας θα πρέπει να πιστεί για την ανάγκη, την αναγκαιότητα αυτών των ε, επιδοτήσεων. Βλέπουμε από τις ε, επιλογές που προτείνει η Κομισιόν, η επιλογή παριθμών 2 είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή προκρίνεται περισσότερο από την Κομισιόν, αυτό νομίζω θα μας οδηγήσει στην καλύτερη κατεύθυνση. Θέλουμε λοιπόν και την ασφάλεια των τροφίμων, θέλουμε όμως συγχρόνως και γεωργούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να εργαστούν και να κερδίσουν με τον ιδρώτα τους το απαραίτητο, ε, την, τα απαραίτητα, το απαραίτητο εισόδημα. Πολλές φορές βλέπουμε ότι έχουμε ένα γεωργό ο οποίος εργάζεται μόνος του στο αγρόκτημά του και κερδίζει 1.500 ευρώ το μήνα για ημέρες των 10 και των 12 ωρών. Ποιος θα ήθελε να δουλέψει κάτω από τέτοιες καταστάσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες. Επομένως, η κλασική εικόνα που έχουμε για τους γεωργούς δεν στέκεται πια αυτό το κλασικό παράδειγμα που είχαμε για τον Γεωργό. Θέλουμε όλοι να υπάρχει καθαρό περιβάλλον. Θέλουμε επίσης οι περιοχές οι οποίες να είναι μειονεκτικές να αντιμετωπίζονται σωστά και να υπάρχει και η προστασία των δημοσίων αγαθών σε αυτές τις περιοχές. Θέλουμε λοιπόν ένα μια ύπεθρο η οποία δίνει δυνατότητες στην ανάπτυξη. Όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολλά. Επομένως, για μένα δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία περίπτωση μια περικοπή του προϋπολογισμού. Ίσα ίσα θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού, τουλάχιστον όμως θα πρέπει να διατηρηθούν τα κονδύλια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Επομένως θα πρέπει έναντι των κυβερνήσεων, έναντι του Συμβουλίου των Υπουργών να κρατήσουμε μια στεναρή στάση και να τους πούμε με τρόπο ο οποίος θα είναι απερίφραστος ότι εμείς στην Ευρώπη δεν μπορούμε να δεχτούμε μια περαιτέρω περικοπή των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά αντίθετα θα πρέπει να βρούμε περισσότερα χρήματα για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Ρόφσκι έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το υπέροχο μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, όπως το περιγράψε ο κ. Μπέρμαν, δεν είναι και τόσο βέβαιο, όμως μπορούμε να φτάσουμε ως εκεί, εφόσον έχουμε την κατάλληλη αγροτική πολιτική διότι χωρίς ε, σοβαρή στήριξη της γεωργικής πολιτικής δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Δεν είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα είναι ο τόπος όπου θα παράγονται τρόφιμα ε, και θα αποστέλλονται έπειτα στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το συζητήσαμε στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου. Στην Αφρική, λόγου χάρη, ε, έχουμε Ινδικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και επενδύουν ψηλά ποσά στην Γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να ε, διασφαλίσουμε ότι θα βρισκόμαστε πάντοτε στην εμπροστοφυλακή της ε, Παραγωγή τροφίμων. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο, είναι δυνατό, αλλά δεν είναι και δεδομένο. Άκουσα επίσης κάποιους συναδέλφους από τους Πρασίνους και την ΚΟΕ να λένε ότι ανησυχούν. Ανησυχούν ότι δεν... μήπως εξασκήσουμε ντάμπινγκ κατά των αναπτυσσόμενων χωρών. Εξ όσων γνωρίζω εγώ συμβαίνει το αντίστροφο. Για παράδειγμα, είχαμε πρόβλημα με τις κατεψυγμένες φράουλες εισαγωγής από την Κίνα ή με το βόηο κρέας ή ε, τα πουλερικά που εισάγαμε από την Βραζιλία και άλλα πολλά προβλήματα αυτού του τύπου. Θα πρέπει λοιπόν να ε, έχουμε υπόψη ότι πολλές φορές πλήττονται δικοί μας οι από τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Έπειτα υπάρχει και το θέμα δεοντολογίας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, ίσο επίπεδο επιδοτήσεων με ανησυχεί σε κάποιο βαθμό όταν κοιτάζω τι πορεία παίρνει η συζήτηση, διότι η διαφορά στο επίπεδο των απευθείας πληρωμών ανεκτάριο είναι τεράστια. Μόνο 500 ευρώ σε κάποιες χώρες και λιγότερο από 100 σε άλλες. Στο σύστημα των επιδοτήσεων λοιπόν Ήταν κατανοητό κάτι τέτοιο. Όμως, ω προ τι πληρωμέ ανεκτάριο, είναι δύσκολο να, δικαι... αιτιολογηθεί. Ε, για μένα είναι απαράδεκτο να αναζητούμε και άλλου λόγου και δικαιολογίε αυτή τη στιγμή για να καλούμε κάτι το οποίο βασίζεται στην ανισότητα να το αποκαλούμε ισότιμο. Είναι άδικο να εικάζουμε ότι οι εύποροι θα πρέπει να διατηρούν τα, τα όσα έχουν και να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον και οι υπόλοιποι να εξακολουθήσουν στην ίδια πορεία. Αυτό δεν είναι ισότητα. Πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε σοβαρές προσπάθειες για να εξεύρουμε λύσεις χωρίς να βλάψουμε τους γεωργούς των παλαιών κρατών μελών και προκειμένου να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Διότι εάν αυτές οι διαφορές παραμένουν θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα. Επίσης μερικές παρατηρήσεις όταν συζητήσαμε για τη συνθήκη τη Λισαβόνα, θυμάμαι ότι όλοι ήταν υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Προσέγγιση. Τώρα, όταν συζητάμε τον προπολογισμό, το ευρωπαϊκό πνεύμα εξανεμίζεται. Δεν υπάρχει πλέον. Μιλάμε για ένα προπολογισμό που είναι κάτω του 1% του 1% του ΑΕΠ. Ε, Πώ λοιπόν αυτό συμβαδίζει με τα μεγάλα ιδεώδη που συζητήσαμε πρόσφατα. Ευχαριστώ. Thank ε, Η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια γενική παρατήρηση και επίσης ένα σχόλιο για την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Η πλειοψηφία των θεμάτων που τέθηκαν από τους συναδέλφους εδώ δείχνουν ότι η ευθύνη μας ως πολιτικών για την ψηφιστική ασφάλεια είναι ένα είδος ευθύνης που δεν μπορούμε πλέον να το αμελούμε. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Ο κ. Σικέρσκι προλίγου είπε ότι τα τρόφιμα είναι θέμα υγείας, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης. Αν δεν φάει κανείς, πεθαίνει. Μην το ξεχνάμε και αυτό σε αυτήν την ε, χρονική περίοδο που έχουμε συστηματική προμήθεια τροφίμων τα πράγματα δεν ε, είναι δύσκολα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Η επισητιστική ασφάλεια προ την πισότητα και την ποιότητα είναι κάτι που διαρκώς πρέπει να το εξασφαλίζουμε. Είναι καθήκον μας. Επίσης θα ήθελα το θέμα αυτό να ληφθεί υπόψη και στην έκθεσή μας, δηλαδή οι συσχετισμοί μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Οι γεωργοί δεν ε, δραστηριοποιούνται σε έναν ιδανικό κόσμο. Ζουν στις περιοχές της Υπέθρου. Η Υπεθρός βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη, ώστε να μην κατοικούν εκεί μόνον γεωργοί, Υπάρχουν και άλλε επαγγελματικέ ομάδε στην Ήπεθρο. Ωστόσο, η ποιότητα διαβίωση των γεωργών σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ποιότητα ε, και την κατάσταση των περιοχών της Υπέθρου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι είναι σημαντικές οι υποδομές στην Ήπεθρο σημαντικές για την γεωργία, για να είναι η γεωργία ανταγωνιστική και για να μπορεί να παρέχει την ποιότητα αυτή διαβίωση που θέλουμε. Θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση σε υπηρεσίε και εκπαίδευση και υγειονομικέ και όλα αυτά είναι αρμοδιότητες της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν να συζητούμε όλες αυτές τις ρεαλιστικές διαστάσεις από κοινού και κάτι άλλο που θα πρέπει να αποσαφηνίσει η δική μας Επιτροπή είναι το εξής. Μιλάμε για την ε, λεγόμενη ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονομική κρίση. Αυτό που έχει προκύψει είναι το εξή. Έχουμε κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον τομέα της γεωργίας. Το 2009 αυτά τα χρήματα επρόκειτο να αποδοθούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης. Ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων λοιπόν θα βελτίωναν τις υποδομές στις περιοχές της υπαίθρου, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν το εξετάσουμε το θέμα αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε ένα βαθμό λειτουργήσε και άσχετα αν ήταν καλή ιδέα ή όχι, θα πρέπει να επαναλάβουμε τις προσπάθειες στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες από την Επιτροπή και να μπορούμε να επεξεργαστούμε επακριβώς την έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Ε. Σας ευχαριστώ. Ο Ζωζε Μανουέλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μία διαπίστωση καταρχήν, η στρατηγική της Ευρώπης 2020 θα πρέπει, θα έπρεπε να συμπεριλάβει και αλλαγές στη γεωργία. Και τώρα μιλάμε για προσαρμογή της γεωργίας στην Ευρώπη 2020, η οποία θα έπρεπε ήδη από την αρχή να έχει συμπεριλάβει πλήρω τη γεωργία σαν κάτι το οποίο είναι κεφαλαιόδε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούσε να είχε εξασφαλίσει την κοινή αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το θέμα της μεθοδολογίας που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τον καθορισμό των κονδυλίων στη γεωργία. Ο κίνδυνος είναι να έχουμε ένα προϋπολογισμό ο θα είναι ο ίδιος ή λιγότερος από ό,τι στο παρελθόν και στη συνέχεια να δώσουμε ένα τμήμα αυτού του προπολογισμού για την πολιτική συνοχή, ένα άλλο για την ε, Ευρώπη 2020 και ένα άλλο κομμάτι για την, για την αγροτική πολιτική. Αλλά η πολιτική συνοχή και η αγροτική πολιτική έχουν ένα σαφές παρελθόν. Έχουν κάποιες δυσκολίες, είχαν όμως και κάποιες επιτυχίες. Επομένως, πρέπει να έχουμε και ένα βασικό επίπεδο εκκίνησης, το οποίο θα είναι το ιστορικό αυτό επίπεδο της ε, γεωργικής πολιτικής, το οποίο είναι ε, εύκολο να το καθορίσει κανείς, γιατί δεν είναι μια καινούρια πολιτική, γεωργική πολιτική. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα αυτού του χρηματοοικονομικού πλαισίου και πρέπει να έχει τα στοιχεία της συνέχειας αυτή η πολιτική για να μην υπάρχουν προβλήματα εκκίνησης στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και καθυστέρηση στην εκταμίευση των ε, ποσών αυτών και μόνο στο τέλος να προσπαθούμε να προλάβουμε τον χαμένο χρόνο. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της ε, Προβληματική τη χρηματοδότηση δεν είναι μονάχα η κλιματική αλλαγή την οποία συζήτησαν ορισμένοι ήδη, αλλά και το θέμα των συνεπειών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να σκεφτούμε πόσα θα πρέπει να είναι τα κονδύλια τα οποία θα μπορέσουν να προλάβουν περαιτέρω φυσικές καταστροφές που μπορεί να είναι σημαντικό το κόστος της πρόληψής τους, αλλά που σίγουρα το κόστος θεραπείας τους είναι πολλαπλό και είναι τεράστιες οι ζημίες οι οποίες ε, θίγουν τους γεωργούς και τους οδηγούν πολλές φορές στη χρεοκοπία. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική την πρόληψη των καταστροφών που μπορούν να πλήξουν τη γεωργία και πώς θα δώσουμε την κατάλληλη υποστήριξη στου γεωργούς μετά από αυτέ τι καταστροφέ, δεδομένου ότι το Ταμείο αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών δεν αντιμετωπίζει τι ανάγκε των γεωργών στο πλαίσιο αυτό. Η Κίνγκα Γκένσου έχει τώρα το λόγο. Ε, ε, ε, κοιτάξτε, Αναφερθήκαμε σε όλα τα στοιχεία της στρατηγικής του 2020. Νομίζω όμως ότι, θα, ότι δεν αναφερθήκαμε τόσο πολύ ε, στο θέμα του inclusive growth, όπως θα το χαρακτήραζε. Πριν και μετά την κρίση, ελπίζουμε μετά την κρίση, δηλαδή μετά από κάποια χρόνια, η απασχόληση θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολούν την Ευρώπη. Και αν ε, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την απασχολησιμότητα στις ε, γεωργικές ε, περιοχές, τότε νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε αργότερα. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της, της συμπερίληψης στην κοινή γεωργική πολιτική είναι πολύ σημαντικό. Εξάλλου και η συνοχή, η περιφερειακή, όχι μόνο η κοινωνική. Αυτό το έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει άμεση σχέση με την ε, περιφερειακή συνοχή. Επίσης αναφέρθηκε ότι η εθνικοποίηση της ΚΑΠ νομίζω ότι ε, αυτή θα ενίσχυε τις ε, διαφορές τα όξινε τις διαφορές και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το τρέχον επίπεδο κονδυλίων. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό. Και θα ήθελα να φέρω και άλλα δύο στοιχεία. Το ένα που αναφέρεται εδώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, πιο δίκαιη κατανομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη να εξισορροπηθούν οι διαφορές ανάμεσα στα παλαιά και τα νεότερα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για λόγους ανταγωνιστικότητας αλλά και εξυγχρονισμού της ε, γεωργίας ε, και είναι σημαντικό ε, για να γίνει η καταστή γεωργία ανταγωνιστικότερη στα νέα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι η μεγαλύτερη διάρκεια και η συνέχεια. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε πολιτική και τρόπους χρηματοδότησης κάθε πέντε χρόνια. Εφόσον μιλάμε για τη διάρκεια των πολιτικών, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά ακριβώς τα στοιχεία της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χρειάστηκε να μιλήσω με τον κύριο Επίτροπο έξω μια στιγμή, συγγνώμη που έλειψα, αλλά σαν εισηγητής για το Αγροτικό Ταμείο μέχρι το χρονικό διάστημα του 2013 θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις για ορισμένα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ πέρα. Αναφέρθηκε το θέμα των πληρωμών που είναι διαφοροποιημένες ανάλογα με τα κράτη-μέλη συζητάμε πάντα για το έτος 2008-2009 αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα είναι τα πράγματα το 2013 και για τα νέα κράτη-μέλη. Γιατί τα παλαιά κράτη ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν νέα κράτη όπως είναι τα βαλτικά κράτη και χώρες όπως η Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αν κοιτάξουμε εδώ πέρα τον πρώτο πυλώνα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ παλαιών και κρατών μελών της διεύνησης. Αν δούμε τώρα τα στοιχεία που αναφέρονται στην ε, σελίδα 7 βλέπουμε ότι κάποιες ε, διαφορές έχουν συρρυκνωθεί. Αν δούμε και τους δύο πυλώνες μαζί και αυτά τα οποία καταβάλλονται τερικά στους γεωργούς. Εγώ στην έκθεσή μου θέλω να εξασφαλίσω μια περαιτέρω μείωση αυτή τη διαφορά. Αλλά αυτό το οποίο με εξέπληξε ήταν ότι μετά από συζητήσει με άλλου συναδέλφου, με υπουργού γεωργίας σε διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βλέπω να υπάρχουν μεγάλε τεράστιε διαφορέ μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη, όχι μεταξύ κρατών μελών. Αυτό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματικής στην ε, Ιταλία μπορεί να έχουμε επιδοτήσεις οι οποίες ποικίλουν από το 1 ως το 10 και στη Γαλλία σε ό,τι αφορά την κατά εκτάριο επιδότηση. Και αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θέλουμε μονάχα δικαιοσύνη μεταξύ κρατών μελών, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Και δεν πρέπει στο μέλλον να υπάρχει μεγαλύτερη ψαλίδα στο εσωτερικό μιας χώρας από ότι μεταξύ διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα το αντιμετωπίσω στην έκθεσή μου και δεν ήξερα ότι ήταν τόσο μεγάλες οι διαφορές γιατί στη Γερμανία μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατηδίων ήταν πολύ μικρές οι διαφορές και ήλπιζα ότι και σε άλλες χώρες είναι το ίδιο αλλά δεν είναι αυτό αλήθεια. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του να υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να δικαιολογήσουμε έναντι τη κοινή γνώμη τι επιδοτήσει αυτέ που δίνουμε στου γεωργού. Στη Βαβαρία υπάρχουν πολλοί γεωργοί. Όπως ξέρετε είναι μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έλαβε χώρα η λεγόμενη μελέτη Μίλεντόρφερ. Και τότε αναφέρθηκε ότι η συνολική αξία της παραγωγής είναι 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο κύριος Μίλεντόρφερ από την Αυστρία ήταν επιφορτισμένος με το να αντιμετωπίσει το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος και την σημασία που έχει η εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης, οι υπόλοιπες σε πάση περιπτώσει παροχές που έχουν να κάνουν με τη γεωργία και οι οποίες δεν πληρώνονται, δεν έχουν κάποιο αντίτιμο με τα ε, με την πώληση αγροτικών προϊόντων. Και είπε ότι έναντι αυτών των 7 δισεκατομμύριων που είναι η αξία της αγροτικής πολιτικής μπορεί να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία η οποία είναι της τάξεως των 3 ε, δισεκατομμυρίων και μόνο ένα 0,5% από αυτήν την ε, παροχή δίνεται αντισταθμίζεται κάποιο τρόπο από τις κρατικές ή τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Επομένως υπάρχει αυτή η προσθέμενη αξία που δίδεται από την ε, γεωργία και η οποία πρέπει να καλυφθεί από τον φορολογούμενο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στην έκθεσή μας. Ότι οι παροχές οι οποίες δίδονται από τους ε, γεωργούς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εδώ πέρα δεν υπάρχει βέβαια δυνατότητα μιας απόλυτης ισοδίκαιας μεταχείρισης. Εδώ ξέρουμε ότι ακόμα και στην, στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης δεν υπάρχει απόλυτη ισοδίκαια αντιμετώπιση, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά και να τονίσουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι παροχές που δίδονται από τους γεωργούς για το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει πολύ σημαντικό τίμημα για τα αγροτικά προϊόντα. Επομένως τα χρήματα που δίνουμε στη Γεωργία δεν τα δίνουμε μονάχα για τους γεωργούς. Τα δίνουμε για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη πίεση προς τους γεωργούς ενώ δεν έχουν την αντίστοιχη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές άλλες εισοδηματικές ομάδες και επαγγελματικέ ομάδες που έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα στην ε, Γερμανία έχουμε 5 εκατομμύρια ανέργους και κοστίζει περισσότερο αυτή η ανεργία από ότι όλος είχαμε μάλλον 5 εκατομμύρια ανέργους και κοστίζει πολύ περισσότερο, τόσο πολύ περισσότερο από ότι όλος ο πρώτος πυλώνας της γεωργίας. Επομένως, θα πρέπει, όπως είπε και ο κ. Σπέκε, να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν καταστρέφουμε πια τη γεωργία των αναπτυσσιωμένων χωρών με τη δική μας γεωργία. Μπορεί αυτό να ίσχυε πριν από 20 χρόνια, αλλά τώρα πια έχουμε καταργήσει τις αγροτικές τις επιδοτήσεις στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Και όπως ελέγχθη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της από τις αγροτικές εξαγωγές της Αφρικής καλύπτει, μόνο, καλύπτει μόνη της τα 80%. Εμείς λοιπόν πολύ περισσότερο από άλλες περιοχές που παράγουν αγροτικά προϊόντα στην, ε, στον κόσμο, εμείς εισάγουμε πολύ περισσότερα προϊόντα. Είμαστε λοιπόν οι πιο ανοιχτοί περιοχή παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αν συγκριθούμε με τι ΗΠΑ χάρη, ή τη Νότια Αμερική. Και δεν υπάρχει ουσιαστικά δασμολογικό εμπόδιο σε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ήθελα λοιπόν να τα αναφέρω. Και τέλος, εγώ προσπαθώ να συντάξω μια έκθεση η οποία θα έχει σαν στόχο να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο δικός μας τώρα εισηγητής από την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και πιστεύω ότι και η δική του έκθεση ελπίζω ότι θα μπορέσει και αυτή να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση μεταξύ μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και αυτή είναι η δική μου ελπίδα να μπορέσω να εξασφαλίσω μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, είναι σχεδόν αδύνατο να συνοψίσω τις τόσο σημαντικές συνεισφορές όλων των συναδέλφων σε αυτή την ευρεία συζήτηση. Μία από τις πρώτες εμπειρίες λοιπόν που είχαμε στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, είναι ότι ήδη μετά από τις 11 το πρωί αρχίζει να μειώνεται ο αριθμός των βουλευτών στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πραγματικά μια μαζική παρουσία όλων των βουλευτών και επομένως δεν μπορώ και εγώ να κάνω μια παρουσίαση συμπερασμάτων εναντίον όλων. Το πιο σημαντικό πάντως είναι να γίνονται αυτές οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των βουλευτών γιατί στη συνέχεια και η γραμματεία της Επιτροπής μας και εγώ ίδιος θα μπορέσουμε να τους δώσουμε μια τέτοια μορφή που να μπορούν να παρουσιαστούν σε όλους τους συναδέλφους και να υπάρξει συζήτηση επί αυτών. Ξεκινώ λοιπόν με αυτό που έλεγε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14 εκατομμύρια γεωργών που διατηρούν ουσιαστικά την ε, οικονομική δραστηριότητα σε περίπου το μισό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές αντιμετωπίζουν διαφορές όχι μονάχα στο πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μέσα στην ίδια την χώρα τους. Και οι περισσότεροι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνουν ούτε καν αυτή τη μέση επιδότηση των 270 ευρώ όπως ανέφερε ο κύριος Ντες. Όταν μιλάμε λοιπόν για ισοδίκαια αντιμετώπιση για να διατηρήσουν το μισό του, της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα 14 εκατομμύρια γεωργών παίρνουν ένα ελάχιστο ποσό επιδότησης. Και εξάλλου έχουμε προδιαγραφές και απαιτήσει ποιότητο και προστασία του περιβάλλοντο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια που είναι πολύ υπέρτερε από αυτέ που ισχύουν σε άλλε περιοχέ του κόσμου που παράγουν επίση αγροτικά προϊόντα. Επομένως μία από τι πρώτε διαπιστώσει στην Επιτροπή μας, η πρώτη, μια από τις πρώτες διαπιστώσεις είναι ότι όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα στο τοπίο της αγροτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι θα θέλαμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάπως εντυπωσιακά διαφορετικές απόψεις και είναι πολύ χρήσιμη μια τέτοια συζήτηση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βρίσκονται οι διαφορές απόψεων. Ο κύριος Επίτροπος νομίζω ότι ήταν αρκετά επικοδομητικός και εγώ τονίζω μερικές από τις πιο σημαντικές δηλώσεις του κυρίου Επιτρόπου, οι οποίες θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην τελική μας έκθεση σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές. Είπε καταρχήν ο κύριος Επίτροπος ότι το κόστος της μη Ευρώπης όπως και στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και στην αγροτική πολιτική. Τι θα κόστιζε στην Ευρώπη να μην έχει μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη κοινή αγροτική πολιτική στο μέλλον. Και τόνισε ακριβώς τι θα σήμαινε αυτό για τα ράφια των σούπερ μάρκετς. Τόνισε ότι η τροφιμική ασφάλεια απαιτεί μια επαρκή χρηματοδότηση της αγροτικής πολιτικής, όπου δεν ισχύει ο κανόνας του ότι το φτηνότερο είναι καλύτερο. Βλέπουμε τι έγινε με τα κινέζικα προϊόντα, τα οποία είναι όσο το δυνατότερο φτηνότερα, αλλά όχι με ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα. Και αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για την ε, διατροφή των Ευρωπαίων πολιτών. Κάνει από τα μέλη της Επιτροπής μας δεν θα ήθελε να αγοράσει μόνο τα πιο φτηνά προϊόντα για την οικογένειά του. Επομένω, η ποιότητα και η ασφάλεια της τροφοδοσίας έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πώς έχουν τροποποιηθεί και οι αγροτικές πρακτικές και η καινοτομία στα πλαίσια των τελευταίων ετών χάρη στη δράση της αγοράς. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να υπάρξει είναι να υπάρξει αντιπαράθεση με για τους περιορισμένους πόρους του προϋπολογισμού μέσα στον ίδιο τον προϋπολογισμό. Θα ήταν ένα πολύ σοβαρό σφάλμα από την πλευρά των μελών της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ εάν δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει ε, συζήτηση για το αν θέλουμε λιγότερη ή περισσότερη γεωργία, λιγότερη ή περισσότερη παιδεία κτλ. Μια τέτοια συζήτηση αυτό οδηγεί σε άμεσες αδικοπραξίες κατά των αντιστοίχων τομέων αυτών του προπολογισμού. Για μας το κύριο εργαλείο ανάλυση, το αναλυτικό εργαλείο που έχουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα πρέπει να είναι η κατανομή των πόρων στις επόμενες χρηματοοικονομικές δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Αυτός πρέπει να είναι και ο γνώμονας που θα ακολουθήσουμε και από την πλευρά αυτή η προσθέμενη αξία για τους γεωργούς και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πέραν οποιασδήποτε διαφωνίας. Είναι κάτι το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Πρέπει λοιπόν στη χειρότερη περίπτωση να διατηρήσουμε τον προπολογισμό γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στρατηγική 2020 Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων των συναδέλφων και του κυρίου Επιτρόπου επίσης είναι ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτημένη γεωργική πολιτική είναι το καλύτερο εργαλείο για να μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική 2020 για την Ευρώπη. Γιατί οι στόχοι αυτή της στρατηγική, τόσο σε θέματα απασχόλησης όσο και σε ποιότητα του περιβάλλοντος συνδέονται άμεσα με την διατήρηση μιας κοινοτική γεωργίας η οποία είναι ισχυρή. Η δομή τώρα αυτής της πολιτικής, όπως είπε ο κύριος Επίτροπος, που είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι από αυτά που είπε ο κύριος Επίτροπος στις απαντήσεις του, γίνεται σαφές ότι θέλει να υπάρχει μία ενιαία κατηγορία στις δημοσιονομικές προοπτικές για την γεωργία. Επομένως οι πιο απλοϊκές ίσως προτάσεις που είχαμε για την μελλοντική διάρθρωση των ε, δημοσιονομικών προοπτικών, δηλαδή εσωτερικές πολιτικές, εξωτερικές πολιτικές και διοικητικές ταπάνες, φαίνεται ότι δεν καλύπτουν αυτή την ανάγκη γιατί ούτε συμπεριλαμβάνουν τις κατευθύνσεις στρατηγικής 2020, ούτε, την, ε, ούτε καλύπτουν την θέληση πολλών συναδέλφων να έχουν μια χωριστή κατηγορία για τους φυσικούς πόρους και διατήρηση των φυσικών πόρων όπου περιλαμβάνεται και η γεωργία. Εάν λοιπόν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη περιοχή που να λαμβάνει υπόψη την συνοχή, θα πρέπει πιστεύω να είναι και η αγροτική πολιτική, του Αγροτικό Ταμείο ανάπτυξη εκεί. Μπορεί να είναι αντίον ο κύριος Επίτροπος και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά εδώ υπάρχει το επιχείρημα ότι ακολουθεί χωροταξικά ε, κριτήρια το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ ακολουθεί μόνο οικονομικά κριτήρια το Ταμείο Συνοχής. Λένε πολλοί συνάδελφοι επομένω ότι πρέπει το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συνδέεται όχι με τη συνοχή αλλά με την ε, αγροτική πολιτική. Για την ευελιξία και για το χρονικό, χρονική διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών είναι σαφές ότι οι περιοχές αυτές δαπανών που απο... απαιτούν μια πιο μακροχρόνια και λεπτομεριακή σχεδίαση θα πρέπει να έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια χρο... χρηματο... δημοσιονομικής προοπτικής. Γι' αυτό δεν μας ικανοποιεί η λύση των πέντε ετών. Όπως είπε και ο κύριος Μπέγκε, νομίζω ότι θα πρέπει να συνδέεται η διάρκεια των ε, προοπτικών να συνδέονται με το επίπεδο του προϋπολογισμού. Θα ήταν αυτοκτονικό με ένα μικρό προϋπολογισμό να έχουμε μακροχρόνιες δημοσιονομικές προοπτικές. Και αυτό είναι και ένα μέσο, ένας μοχλός πίεσης στα κρατη ότι δεν μπορούμε να έχουμε ε, σύντομες δημοσιονομικές προοπτικές εάν δεν μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε επαρκή χρηματοδότηση του προϋπολογισμού στο άμεσο μέλλον και είναι απαραίτητο να υπογραμμίσω ενώπιον της Επιτροπής μας ότι αν 80% των δαπανών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στον τομέα της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής γεωργίας, εάν πρέπει αυτές οι δύο πολιτικές να έχουν μεγαλύτερα διαστήματα δημοσιονομικών προοπτικών, είναι λογικό να υπάρχει και σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ευρύτερη, μια μεγαλύτερη χρονικά δημοσιονομική περίοδος. Μεταξύ 7 λοιπόν και 10 ετών. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα πρέπει να το λάβω υπόψη μου, ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι το βλέπουν έτσι. Το θέμα της ευελιξίας, ας είμαστε ειλικρινείς. Είδαμε τι έγινε στο έγγραφο το οποίο παρουσιάσαμε για την ευελιξία στις δημοσιονομικές προοπτικές. Η γεωργία είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει στην ευελιξία. Αυτό το οποίο επέτρεψε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην Κομισιόν και το Συμβούλιο να καλύψει απρόβλεπτες ανάγκες το 2006 ήταν μονάχα το ότι υπήρχαν πλεονάσματα στην αγροτική πολιτική και στην ε, πολιτική αγροτικών θεμάτων. Αυτό δεν είναι ο πιο υγιής τρόπος για να ασκούμε μια πολιτική προϋπολογισμού. Ξέρουμε ότι αυτό όμως έλαβε χώρα μέχρι τώρα. Γι' αυτό ένα από τα πιο αμφίμαχα σημεία τα οποία παραμένει για την πρόταση που θα διατυπώσει η Επιτροπή μας είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την ευελιξία στις διάφορες κατηγορίες του προπολογισμού χωρίς να θίγεται η κοινή αγροτική πολιτική που είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε κάνει μέσα στα πλαίσια της τελευταίας περίοδου δημοσιονομικών προοπτικών. Επίσης το θέμα της ε, απλοποίησης το οποίο έθιξε ο κύριος Μπέργκερ. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς κανονισμούς για διαφορετικές περιοχές της κοινή αγροτικής πολιτικής, όπως δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις για διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και θέλουμε και η Επιτροπή και ο κύριος Επίτροπος να δεσμευτούν για την απλοποίηση των διαδικασιών. Όλα αυτά είναι μια σημαντική πρόταση λοιπόν που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε οριζόντιο επίπεδο. Δυστυχώ ο εισηγητής μας, εισηγητή σας δεν μπορεί να περατώσει την εκθεσή του προτού δώσει στη δημοσιότητα και την ανακοίνωσή της η Κομισιόν. Σας λέω και πάλι ότι οι περισσότεροι ομιλητέ ακολούθησαν αυτήν την κατεύθυνση, ήταν σαφές ποιοι ήταν η πλειοψηφία των ομιλητών και στην ειδική μας Επιτροπή και στην Επιτροπή Γεωργίας και θα προσπαθήσω να αποτυπωθούν αυτά στην έκθεσή μου τις επόμενες εβδομάδες <clears throat> ώστε, εάν συμφωνούν οι συντονιστές, να παρουσιαστεί αυτό το έγγραφο που και πάλι στην Επιτροπή μας το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτον για την πειθαρχία που επέδειξαν και δεύτερον βέβαια και για τις παρεμβάσεις τους. Τώρα, αν με ρώταγαν εμένα ε, τι απέδωσε αυτή η συζήτηση, θα το έλεγα πολύ απλά και γρήγορα Δηλαδή εμείς δεν επιθυμούμε επανάσταση όσον αφορά την μελλοντική ΚΑΠ. Θέλουμε μια απλή μεταρρύθμιση που να οδηγήσει στη χρηματοδότηση της ε, παραγωγής ε, δημόσιων αγαθών. Αυτό είναι το ένα. Και δημόσια αγαθά είναι ασφάλεια των ε, τροφίμων, προστασία εδάφους και όλα αυτά τα οποία κατανοεί κανείς κάτω από δημόσια αγαθά. Αυτό πρέπει να κάνουν οι γεωργοί, αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Να... Αυτή είναι η στόχη για το μέλλον. Τώρα, ε, τα κονδύλια που υπάρχουν πρέπει να κατανέμονται δικαιότερα. Και εγώ ε, τώρα το από τον κύριο Ντες. Τώρα τα άκουσα ότι υπάρχουν διαφορές όχι μόνο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και μέσα στο ίδιο το κράτος όσον αφορά το θέμα αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερα κονδύλια από αυτά που μας είχατε διαθέσει κατά το παρελθόν. Αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα. Βέβαια εγώ δεν μπορώ να θεωρηθώ η κορυφή της Γεωργίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αν με ρωτήσει κάποιος κάπου εκεί καταλήξαμε όλοι. Έτσι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς. Βεβαίως γνωρίζω ότι δεν ικανοποιώ όλους με αυτά που είπα. Ε, θέλω να πιστεύω όμως ότι ευχαρίστησα την ε, πλειοψηφία εκείνων που παρενέβησαν. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 3 της ημερήσιας διάταξης. Τώρα θα κάνω εγώ τις ανακοινώσεις μου γρήγορα. Εχθές λοιπόν ε, ε, ακούσατε στις συνεδρίες των συντονιστών, αυτό που ενδιαφέρει είναι η επόμενη συνάντησή μας. Αποφασίσαμε ότι θα καλούμε κάθε φορά τους αρμόδιους επιτρόπους. Είπαμε όμως ότι δεν θέλουμε να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα καθορίζουμε ποιος είναι αρμόδιος. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλέσαμε τον πρόεδρο κύριο Μπαρόζα να μας στέλνει εκείνος τους επιτρόπους. Και το έκανε αυτό. Έστειλε τον κύριο Σόλος ε, για τη γεωργική πολιτική. Την 1η Φεβρουαρίου <clears throat> θα συζητήσουμε για έρευνα και ανάπτυξη, ε, ενέργεια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εκεί λοιπόν ξέρουμε ότι έχει κληθεί η Επίτροπος Αρμόδια για την έρευνα ε, να έρθει εδώ. Επίσης ο κύριος Ότιγκε, αρμόδιος επίτροπος για την ενέργεια και ο επίτροπος κύριος Κάλλας που είναι αρμόδιος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Την ε, οριστική δέσμευση έχουμε μέχρι τώρα μόνο από την Επίτροπο Έρευνας και θα δούμε στη μεθεπόμενη συνεδρίαση στις 10 Φεβρουαρίου εκεί θα ασχοληθούμε με τη συνοχή και την αλληλεγγύη και έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί ότι θα έρθει ο Επίτροπος ε, κύριος Χάν και ο Επίτροπος κύριος Αντόρ Ε, πάμε τώρα πίσω στην 1η ε, Φεβρουαρίου. Ε, Πίτροπος Πίμπαλτς έχει κληθεί, αλλά δεν έχει απαντήσει οριστικά κατά πόσον θα μπορέσει να έρθει. Όσον αφορά στα έγγραφα εργασίας, ο Σαλβαντόρ ήδη τοποθετήθηκε, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο επ' αυτού. Και έχουμε ήδη πει ότι αν διαπιστώσουμε ότι ο χρόνος μας δεν μας φτάνει, θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε μία περαιτέρω συνάντηση για την Επιτροπή μας και το κάναμε αυτό. Ορίσαμε την 5η 10η Μαρτίου. Αυτή είναι η εβδομάδα του Στρασβούργου και θα συνεδριάσουμε το πρωί μέχρι την ώρα των ψηφοφοριών. Εχθές στις συνεδρίες των συντονιστών είπαμε επίσης ότι θέλουμε να αντιδράσουμε στην ερώτηση της διάσκεψης των Προέδρων, οι οποίοι είπαν ότι όλες οι επιτροπές πρέπει να συνεισφέρουν στο ψήφισμα το οποίο θα κατατεθεί στην Εαρινή Σύνοδο εκ μέρου των πολιτικών ομάδων η διάσκεψη των Προέδρων θα συνεισφέρει και αυτή. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα συμβάλλουμε. Από τα έγγραφα εργασίας του Σαλβαντόρ θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια σύντομη περίληψη και να αναφέρουμε όλα αυτά που έχουν υποθεί εδώ για την Ευρώπη 2020 για την ανταγωνιστικότητα. Θα σας το στείλουμε το έγγραφο αυτό και αν έχετε ε, σχόλια τα οποία θα θέλετε οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν θα πρέπει να μας τα στείλετε ε, έχουμε χρόνο μέχρι την επόμενη εβδομάδα μόνο που να πω αυτό που είπα και χτες το βράδυ. Δηλαδή αυτή θα είναι η συνεισφορά μας για τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Η διάσκεψη των Πρόεδρων θα συνοψίσει όλες τις παρεμβάσεις ε, των Επιτροπών και από εκεί θα συνταχθεί το ψήφισμα. Δηλαδή αυτά που θα στείλουμε εμείς δεν θα τα βρούμε όλα ε, κατά γράμμα στην πρόταση του ψηφίσματος, ο καθένας θα πρέπει στην δική του την πολιτική ομάδα, αν κάτι του είναι σημαντικό, να το επισημάνει και να επιμείνει να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο. Αυτή θα είναι η συνεισφορά μας. Ως Επιτροπή πήραμε μία ερώτηση από την Βουλή των Λόρδων της Μεγάλης Βρετανίας οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν έτσι μια εικόνα του τι μορφή θα έχει ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα σε επόμενα έτη. Τίθεται λοιπόν μία σειρά ερωτημάτων και οι Βρετανοί που είναι στη Βουλή των Λόρντων ε, πήραν και αυτοί αυτό το ερώτημα και εμείς βέβαια ως Επιτροπή οι συνάλληλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και εγώ θα προσπαθήσω ως πρόεδρος της Επιτροπής να δώσω μία απάντηση στους Λόρδους. Ε, χτες μάλιστα ε, λέχθηκε το εξής που το βρίσκω πολύ σημαντικό. Οι Λόρδοι επισημαίνουν ότι ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα Και ε, μας ενδιαφέρει και εμά η έκθεσή τους, γιατί αυτή η έκθεση ε, είναι σημαντική για τη δουλειά μας. Και όπως ξέρουμε από το παρελθόν, οποτεδήποτε η Βουλή των Λόρδων ε, έκανε τέτοιου είδου έρευνες, ήταν πολύ καλή η δουλειά τους, ιδιαίτερα αξιόπιστη και πολύτιμη και τα αποτελέσματα των ερευνών τους μπορέσαμε, μπόρεσαν όλα να τα χρησιμοποιήσουν για περαιτέρω έρευνα. Αυτά είχα να πω εγώ ε, ως ανακοινώσεις προέδρου. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφο επιθυμεί να προσθέσει κάτι. κανεί δεν θέλει να πει τίποτα άλλο. Καλή όρεξη. Γεια σα. το καλή όρεξη λέει η πρόεδρο. είναι μία ίσως γερμανική αλλά όχι και μόνο ευχή